να ευχαριστήσω όσους έχουν έρθει και να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Στο σημείο 19, με ιδιαίτερη χαρά, υποδέχομαι τον υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Στη δική μας τη γλώσσα, αυτόν τον οργανισμό τον ονομάζουμε Bilbao, οργανισμό του Bilbao. Αυτό βέβαια δεν αφορά το μέλλον, το, τις μελλοντικές σας αρμοδιότητες. Πάντως με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι σε αυτή την Επιτροπή. Όπως τα ξέρετε φτάνετε σε μια στιγμή που υπό την αιγύδα του κυρίου Τάκαλα και των συναδέλφων του το κοινοβούλιο εδώ έχει συμμετάσχει σε μια μεγάλη προσπάθεια προβολής του έργου των οργανισμών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που έρχεστε σε αυτή τη σημαντική στιγμή, διπλά σημαντική, γιατί το Κοινοβούλιο με εκπρόσωπό του την κυρία Ντελή εξετάζει αυτή τη στιγμή τους κανονισμούς για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. Εκπονούνται αρκετές μελέτες τις οποίες και εμείς τώρα μελετούμε. Έχετε λοιπόν ε, αναλάβει ένα καθήκον πολύ επίκαιρο και σημαντικό. Ο διορισμός σας θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε πολύ άνετα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα, διότι δεν βρίσκεστε εδώ ούτε για να σας εγκρίνουμε, ούτε για να σας απορρίψουμε. Απλώς θα συζητήσουμε θα επικοινωνήσουμε και έτσι μπορείτε να μας παρουσιαστείτε. Και να μας πείτε και ποιο είναι το κληροδότημα που θα σας αφήσει ο κύριος Τάκαλα, τον οποίο θα χαιρετήσουμε στο τέλος της συνάντησής μας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα και ελπίζω να μπορέσω να συμμετάσχω σε αυτές τις συνεδριάσεις αρκετές φορές στο μέλλον. Ενημερώθηκα ότι έχετε λάβει το βιογραφικό μου σημείωμα, επομένως θα σας δώσω απλώς μια σύντομη περίληψη για την ε, επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ξεκίνησα ε, στη Γερμανία στην επιθεώρηση εργασίας, κατόπιν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εργάστηκα στην υπηρεσία του Μπιλμπάου για έξι χρόνια και... Ε, τα τελευταία χρόνια ήμουνα επικεφαλής του τμήματος ε, περιβάλλοντος εργασίας. Ε, κατόπιν μετέβη στο Βερολίνο για το Ινστιτούτο Ασφάλειας ε, και Υγείας στον χώρο της εργασίας και κατόπιν έγινα διευθύντρια μιας νέας πρωτοβουλίας η οποία ξεκίνησε με την πρωτοβουλία Νέα Ποιότητα Εργασίας και ε, ιδρύθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας με συνολικό στόχο για περισσότερους και καλύτερους χώρους εργασίας και κοινωνικό διάλογο και ε, εκεί από την εμπειρία μου ως διευθύντρια έχω να σας πω ότι... Ε, καθορίστηκε το σκεπτικό μου και η προσέγγιση που έχω ως προς την εργασία. Βάσει της πείρας μου από τα τελευταία 20 χρόνια, θεωρώ ότι η ασφάλεια στο χώρο της ε, εργασίας και η υγεία έχει κάνει σημαντικές πρόοδους τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε τα στοιχεία και τις επιπτώσεις ε, της πολιτικής μας ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της πολιτικής ιδίως λόγω των δημογραφικών αλλαγών. Οι άνθρωποι γυράσκουν, πρέπει να εργάζονται περισσότερο και ε, να μένουν περισσότερο χρονικό διάστημα υγιείς. Αυτό δεν είναι μόνο ηθική και ανθρώπινη υποχρέωση για να προάγουμε την υγεία, αλλά είναι και οικονομική πλέον ανάγκη. Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουμε πώς ε, είναι η καλή και αξιοπρεπή εργασία. Ε, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που είναι υγιείς και έχουν κίνητρα συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις και επίσης έχουμε βιώσει και το γεγονός ότι η τεχνογνωσία δεν ε, μεταλαμπαδεύεται στο χώρο της εργασίας κατά τρόπον ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν εύκολα οι επιχειρήσεις. Εξακολουθεί λοιπόν να υφίσταται η ανάγκη να πληρώσουμε το κενό μεταξύ των υφιστάμενων γνώσεων και της επαρκούς τους εφαρμογής στις επιχειρήσεις επιχειρήσεις. Βάσει της εμπειρίας μου και των γνώσεών μου, όταν αναφέρομαι σε επιχειρήσεις, ε, σαφώς ε, αναφέρομαι ε, και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομίας και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά την άποψή μου, Τέσσερι είναι οι τομείς που αποτελούν προτεραιότητα όταν προάγουμε την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη και σε αυτούς του τέσσερι τομείς ε, ο οργανισμός μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι γνωρίζετε ήδη ότι είναι ένας από τους βασικούς ε, παράγοντες ε, ο οργανισμός. Καταρχάς θα πρέπει ε, να διαβιβάσουμε το μήνυμα της ασφάλειας και την υγεία στον χώρο της εργασίας και να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια χάρτα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, να υπάρχει κατάλληλη δικτύωση με τις ομάδες στόχο ώστε να αναπτύξουμε και να διαβιβάσουμε πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες ε, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την εργασία και τέταρτον να υπάρχει mainstreaming στην ε, ε, ασφάλεια στον χώρο της εργασίας, δηλαδή ε, να είναι οριζόντιο το θέμα για δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τώρα, πώς βλέπω το ρόλο του οργανισμού. Ο ρόλος του οργανισμού του Μπιλμπάου είναι ζωτικός ε, σε όλους τους τέσσερις τομείς που σας ανέφερα προηγουμένως και ο οργανισμός συνεισφέρει και στους τέσσερις αυτούς τομείς σε στενή συνεργασία με το δίκτυο των οργανισμών, ε, με τη διαβίβαση τεχνογνωσίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεισφέρει στην ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εργασία και ε, μας ενδιαφέρουν ε, επίσης τα όσα γίνονται στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για κληρονομιά του οργανισμού, ένα προσγειωμένο δίκτυο το οποίο βασίζεται και στη στενή συμμετοχή των συνδικάτων και των οργανώσεων των εργοδοτών. Τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός ε, διεξήγαγε με επιτυχία σημαντικά προγράμματα και στοιχεία τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο της εργασίας, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα το οποίο διευκόλυνε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα θέματα αυτά και έχουμε και κάποια στοιχεία πλέον από τις ίδιες επιχειρήσεις για τις ανάγκες τους ε, και το τι χρειάζονται από πλευράς οργανισμού ε, όσον αφορά τις πληροφορίες που μπορεί να τους δώσει. Επίσης υπάρχει και η ενεργός αξιολόγηση κινδύνου. Και επειδή έχω εργαστεί και στο παρελθόν στον οργανισμό, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό μέσο ώστε τα κράτη-μέλη να ε, λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζεται και αυτό ε, αναπτύχθηκε στα κράτη-μέλη ξεκίνησε ως κάτι καινούριο και αναπτύσσεται έτσι περαιτέρω και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ζωτική σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το παράδειγμα όμως καταδεικνύει πώς ε, η εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα. Υπάρχουν ε, ποικιλόμερφα παραδείγματα επιτυχίας ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιούσα στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, μη νομοθετικά μέσα όπως συλλογικέ συμβάσεις ή προγράμματα που βασίζονται σε αυτές τις συλλογικέ συμβάσεις, τα οποία ήταν πολύ επιτυχή ε, επειδή έγιναν και σε στενή συνεργασία με τα συνδικάτα και τις οργανώσεις των εργαζομένων. Η επιθυμία μου είναι και νομίζω ότι ο οργανισμός ούτως ή άλλως βρίσκεται στο σωστό δρόμο, να καθορίσουμε έναν οδικό χάρτη για την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη, ώστε οι ομάδες ε, στόχος να μπορεί να έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα στις πληροφορίες που χρειάζονται. Το δεύτερο, το να διαβιβάσουμε το μήνυμα, αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες εκστρατείες, ε, υπάρχουν εκστρατείες οι οποίες έχουν πάει πολύ πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν από την αξιολόγηση του 2007. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εκστρατεία παγκοσμίω και εγώ προσβλέπω στην προετοιμασία των δύο επόμενων ε, στρατηγικών. Τα πρώτα δύο χρόνια θα είναι ε, αφιερωμένα στην πρόληψη βάσει της εταιρικής σχέσης και επίσης ε, η επόμενη εκστρατεία είναι οι κίνδυνοι από κοινωνική πλευρά που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Επίση, θέλω να προωθήσω και τη συνεργασία με τη φυστάμενα δίκτυα, όπω για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Υγεία στο χώρο τη εργασία ή την Επιτροπή Επιθεωρήσεων Υγεία. Υπάρχει καλή ε, συνεργασία επίσης και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ε, ο νυν διευθυντής θα σας παρουσιάσει και τα όσα γνωρίζει για το θέμα αυτό. Ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ενδυνάμωση και την αναγνώριση κυρίως των νέων ανθρώπων Όσο νωρίτερα ξεκινήσουν, τόσο καλύτερα αντιλαμβάνονται και διαμορφώνουν απόψεις, αυτό το γνωρίζουμε και ο οργανισμός ε, θα συνεργαστεί και με ζωτική σημασία οργανισμούς ε, στο θέμα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Είχαμε ένα σεμινάριο στις 30 Ιουνίου στις Βρυξέλλες όπου συμμετείχαν όλοι οι οργανισμοί, ο οργανισμός του Δουβλίνου, ο οργανισμός Ευρωπαϊκή Ένωση, ο SHE, εμείς ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε. Κάποια στοιχεία τώρα για το ρόλο του Διευθυντή. Γνωρίζω ποια είναι τα καθήκοντα του διευθυντή από τότε που εργαζόμουν στον οργανισμό του Μπιλμπάου, αλλά πλέον Έχω και μια άλλη εικόνα για το ρόλο του Διευθυντή. Είναι σαφές ότι εγώ είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού και είμαι υπόλογη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω φυσικά ποιες είναι οι ευθύνες μου, παραδείγματο χάρη η εφαρμογή του προπολογισμού και η χρηματοοικονομική διαχείριση του οργανισμού βάση του άρθρου 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που ισχύει για το Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο βέβαια διαπιστώνω και πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και φυσικά η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επομένως είναι σαφές για μένα ότι είστε σημαντική εταίροι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει ένα μικρό γραφείο ε, μίας διευθυντού που ε, θα δώσει και τη σαφή ένδειξη ότι προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε, ότι ο οργανισμός δηλαδή θέλει να έχει τακτική και ισχυρή σχέση και με την Επιτροπή σας και τις υπόλοιπες Επιτροπές του Κοινοβουλίου και με άλλους ζωτικής σημασίας εταίρους. Ε, γνωρίζω βέβαια και την ομάδα εργασίου ας για το μέλλον των οργανισμών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευπρόσδεκτα τα όσα έχουν να μας πούν και ξέρω ότι οι αξιολογήσεις αυτές είναι ο λογικός τρόπος να εξετάσουμε μια κατάσταση εξετάζονται ε, τα στοιχεία από διάφορες οπτικές γωνίες και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και για τη μελλοντική προστιθέμενη αξία του οργανισμού και θα δούμε φυσικά και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν για τους οργανισμούς εν γέννη. Είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως σε όλους τους οργανισμούς και τα δίκτυα άλλωστε. Ο οργανισμός μας ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Εγώ εργάστηκα στον οργανισμό για πάνω από 5 χρόνια. Έχω εργαστεί και εκτός οργανισμού ως ε, ε, συνεταίρος για πολλά χρόνια και φυσικά ήδη έχω κάποιες ε, προτάσεις αλλαγών και βελτιώσεων Γνωρίζετε την εμπειρογνωμοσύνη μου, γνωρίζετε το βιογραφικό μου και την εμπειρία που αποκόμισα τα τελευταία 20 χρόνια. Θα ήθελα ίσως να επισημάνω ότι ό,τι κάνω και ό,τι θα κάνω ως Διευθύντρια θα βασίζεται στην ισχυρή βούλησή μου η ασφάλεια και η υγεία στον χώρο της εργασίας να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέρα έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γυράσκουσα κοινωνία, το γεγονός ότι ε, υπάρχει κόστος από 1 3% του ΑΕΠ, το κόστος των ατυχημάτων, ε, τα προβλήματα που δημιουργούνται σε ανθρώπινο επίπεδο και φυσικά και το κόστος της υγείας. Όλα αυτά εξαρτάται από το γεγονός ε, ότι το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί. Και επίσης κάτι που είπα και στην αρχή, ότι θέλουμε να προχωρήσουμε δηλαδή και στην Ευρώπη αλλά και εκτός συνόρων, Έχουμε για παράδειγμα τις καναδικές δραστηριότητες ε, που ξεκινούν κάποια πράγματα ε, για τον αμίαντο και θα πρέπει να σας πω ότι είναι κρίμα γιατί πριν από 20 χρόνια συμμετείχα στην Αυστρία στην απαγόρευση της χρήσης αμιάντου και για μένα ήταν μια πολύ επιτυχής μέρα η μέρα που ο υπουργό υπέγραψε την απαγόρευση του αμιάντου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινωνία που θα πρέπει να δείξει ε, υπευθυνότητα στις δράσεις του Καναδά και θεωρώ ότι και ο οργανισμός έχει ευθύνη και θα πρέπει να υποστηρίξει ε, αυτές τις διαδικασίες. Ελπίζω να τήρησα και το χρονικό διάστημα που μου δώσατε. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε για την ε, ενθαρρυντική αυτή παρουσίαση. Η κυρία Αντελή θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Να σας ευχαριστήσω κύριε Σάντριτσκα που είστε μαζί μας. Ο οργανισμός του Μπελμπάο που είχα την τύχη να επισκεφθώ μαζί με τα μέλη της αντιπροσωπείας ε, επιτελεί ένα έργο που δεν είναι καθόλου αρκετά επαρκώς γνωστό. Για μένα και για όλους εμάς τους βουλευτές και στα πλαίσια της έκθεσης για τις συνθήκες ασφάλειας και γενής στο χώρο εργασίας είναι πηγή λοιπόν πολλών χρήσιμων ε, πληροφοριών. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δούμε το θέμα αυτό κατά τρόπο συνολικό. Είναι ένα ζήτημα που δεν έχει μόνο διαστάσεις ανταγωνιστικότητας, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποφύγουμε τα ανθρώπινα δράματα, τα ανθρώπινα θύματα, τα θανατηφόρα ατυχήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας θέσω το εξής ερώτημα. Σήμερα Μπορώ, Πρόεδρε, να πέρασω από αυτές τις ερωτήσεις. Ωραία. Να σας ρωτήσω ποια είναι για σας, ποιος είναι ο συσχετισμός μεταξύ υγείας ασφάλειας και διάρκειας του χρόνου εργασίας. Επίσης, τις συνθήκες υγείας πώς τις αντιμετωπίζετε για τα νέα επαγγέλματα. Αγαπητοί συνάδελφε, μπορείτε να θέσετε όσα ερωτήματα θέλετε. Απλώς να σας θυμίσω ότι η κυρία Σλάτερσεκ είναι υποψήφια, υποψήφια για τη θέση του διευθυντή. Είναι διευθύντρια. Στον οργανισμό αυτό Οπότε καλό θα είναι να τη θέσετε ερωτήματα για θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά της. Κοιτάξτε, το θέμα που θα ήθελα να μου διευκρινίσει είναι ο χρόνος εργασία και ο σχετισμό με την, με την υγεία και την ε, ασφάλεια. Επίσης, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο φάσμα διαφορετικών ε, προγραμμάτων, η απόκληση δηλαδή των ευρωπαϊκών οδηγιών με τα εθνικά προγράμματα. ως προς την ενημέρωση δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε και ω προ την ανταλλαγή των πληροφοριών εμπειρικά και πειραματικά. Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία από διάφορε χώρε που δεν είναι γνωστά στου υπόλοιπου. Ευχαριστούμε, ο κύριο Σέρκα. Και μετά, κυρία Στάνγκλουκ. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να καλωσορίσω την κυρία Σετ Λάσερ, αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ε, είναι αδύνατο για μένα, γιατί είναι στα γερμανικά, παρόλο που αντιμετωπίζω και πολύ πιο δύσκολα ονόματα στη χώρα των Βάσκων. Και να αποχαιρετήσω τον κύριο Τάκαλα, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ε, μας αφήνει πολύ καλές αναμνήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το δικό σας το έργο γίνεται πολύ δύσκολο, διότι πρέπει να βελτιώσετε τα πράγματα μετά από κάποιον ο οποίος ήταν άριστος. Ε, δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, αν και μετά από όσα άκουσα από πλευρά σας, νομίζω ότι έχετε τις δεξιότητες ε, και τη βούληση και τις ανάλογες δεσμεύσεις έχετε αναλάβει για να προχωρήσετε το ζήτημα. Επομένως, έχετε το πράσινο φως από πλευρά μας. Ε, είναι η μέρα λοιπόν που σας καλωσορίζουμε και θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση. Τη ρώτησε βέβαια κυρία Ντελή ε, και η πρόεδρος είπε να μην ρωτήσει. Δεν θα ρωτήσω λοιπόν και εγώ τίποτα σήμερα. Κάποιες σκέψεις μόνο να πω. Σήμερα θα δούμε πώς η Επιτροπή Απασχόλησης θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του έργου μας ε, το θέμα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Είστε παρούσα, θα συζητήσουμε τη στρατηγική 2007-2012, θα δεχθούμε τους φίλους από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τμήμα των δεσμεύσεών μας και εσείς ε, κυρία μου θα πρέπει εδώ στην Επιτροπή Απασχόληση θα βρείτε τους καλύτερους συμμάχους σας. Βέβαια μπορούμε να γίνουμε και ο χειρότερός σας εφιάλτη ε, θα πρέπει ε, να δούμε και τι κάνουν αυτοί που δεν τους αρέσει η Ευρώπη. Όχι δεν τους αρέσετε εσείς, αλλά δεν τους αρέσει η Ευρώπη. Οπότε μπορεί να υπάρξει και αντικείμενο επίθεσης, διότι υπάρχουν οι που είναι κατά της Ευρώπης. Εδώ όμως, στην Επιτροπή μας, η πλειονότητα εκτιμά ιδιαίτερα τη σημασία του οργανισμού και ε, το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν συλλογικές απαντήσεις ε, απαντήσεις που δεν θα είναι ατομικές, αλλά θα είναι απαντήσεις της κοινωνίας, ώστε να έχουμε πρόληψη και επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που δημιουργούν ε, τα καθημερινά δράματα των ανθρώπων, τα ατυχήματα στο χώρο της εργασίας ε, ε, και όλα όσα σχετίζονται με την υγεία. Για μας είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει πρόληψη, να υπάρχουν μελέτες, να γνωρίζουμε, να ανταλλάσσουμε τις βαλτιστές εμπειρίες και να δίνουμε το δέον δυναμικό στην κοινωνία και να υπάρχουν νέες ιδέες που είναι επίσης σημαντικό, διότι αν αφήσουμε στην αγορά τα θέματα και τα θέματα του, μεγαλύτερου δηλατού κέρδους θα ξεχάσουμε την πρόληψη. Εσείς το είπατε, γιατί εργάζεστε πολύ, πολλά χρόνια στον οργανισμό, ε, ότι ο οργανισμός έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία. Εγώ προήλθα από μια χώρα που δεν ήταν ε, από τους πρώτους, ήρθε το 1986 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα μου ήταν μεγάλη σημασία. Ο οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές πρακτικές, οι οποίες μας επέτρεψαν σε λίγα χρόνια να φτάσουμε στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της γνώσης που είχαν οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δυστυχώ δεν μπαίνει στην οτροπία των λογιστών που ελέγχουν τον οίκο μα, αλλά εμεί που είμαστε ευρωβουλευτέ και εργαζόμαστε εδώ κατανοούμε αυτά τα πράγματα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε ακόμα καλύτερα. Διάβασα τι προτεραιότητε, σα, δεν πρόκειται να πω τίποτα, συμφωνώ με τα όσα λέτε για το ρόλο του Διευθυντή. Έχουμε αναλάβει μια δέσμευση, διότι εμένα με εντυπωσίασε και ένα σεμινάριο που κάναμε πολύ πρόσφατα για το θέμα του αμιάτου. Νομίζαμε ότι είχε επιληθεί το ζήτημα, αλλά τελικώς δεν έχει επιληθεί και τα στοιχεία είναι θεαματικά και είναι και πονίδιστα. Πρόκειται για μία μάστιγα η οποία συνεχίζεται και ακόμα δεν γνωρίζουμε σε τι ποιότητα και σε τι ποσότητα υπάρχει ο αμύαντος, διότι δεν έχουμε καλά στατιστικά στοιχεία για όλα τα ε, κτίρια τα οποία έχουν ε, ε, πληχθεί και για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σε συνθήκες κινδύνου. Εγώ σας ζητώ να κάνετε μεγάλες προσπάθειες, διότι υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία πολύ σημαντικά για τους ανθρώπους που συνεχίζουν να εργάζονται εκεί και τα προβλήματα που δημιουργεί και δημιούργησε στο παρελθόν είναι πολύ σημαντικά. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ελπίζω να συνεργαστούμε στο μέλλον ε, ε, για την επίλυσή του. Κύριε Στέμπλοκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Σέτλατσεκ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρουσιαστήκατε εδώ και τόσο αναλυτικά και από όσα άκουσα μόλις τώρα είμαι σίγουρη ότι η συνεργασία μαζί θα είναι εξίσου καλή όπως και με τον κύριο Τάκαλα. Η υπηρεσία του Πιλμπάου είναι πάρα πολύ σημαντική για τη δική μας εργασία. Δύο φορές έχω πάει ήδη και γύρισα με πολύ καλές ιδέες και ναύσματα που προέρχονται από τις έρευνες και την παρουσίαση της υπηρεσίας αυτής. Στην παρουσίασή σας ε, αναφερθήκατε στις κύριες προκλήσεις και χάρηκα ότι άκουσα ότι θέλετε να τοποθετήσετε τον άνθρωπο στο επίκεντρο και να υπάρχει καλή και αξιοπρεπή εργασία, ότι κοιτάμε δηλαδή τον άνθρωπο, πράγμα που δεν πραγματοποιείται πάντα στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά την μέχρι τούδε εργασία σας ως ε, ε διευθύντρια της πρωτοβουλίας για την καλύτερη ανθρώπινη ποιότητα της εργασίας. Βλέπετε να υπάρχει κάποια δυνατότητα να πάρετε αυτά, αυτές τις εμπειρίες και να τις μεταφέρετε στην υπηρεσία του Μπιλμπάου. Ιζαβετ Λίνγκ, ο πρόεδρος. Και μετά Ντανούτα ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την επιτροπή όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Τάκαλα για το έργο που έχει επιτελέσει στο παρελθόν. Είχαμε πάρα πολύ υποκοδομητικές ερωτήσεις μαζί σας ε, καθ' όλη τη διάρκεια που ήσασταν διευθυντής και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά που έχετε επιτελέσει και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και πολύ καρποφόρες συζητήσεις και στο μέλλον. Αναφερθήκατε σε προληπτική προστασία της υγείας ε, και της ασφάλειας. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη αξιολόγηση κινδύνου για τις ΜΜΕ. Είναι πολύ χρήσιμο και εσείς είπατε ότι έχει προχωρήσει περισσότερο ή θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο. Αν έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού θα ήταν χρήσιμο. Και αναφερόμενοι σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ε, το έργο που επιτελείται έχει ευρύ ακροατήριο, γιατί ίσως είστε γνωστοί εδώ, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν καθόλου τι κάνει η υπηρεσία του Μπιλμπάου. Και ίσως ε, έχει φτάσει πια η ώρα να αναγνωρίσουν όλοι πόσο σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται εκεί. Και αναφερόμαστε σε αυτά που είπε ο κύριος Σέρκας για τον Αμίαντο, θα μπορούσα πραγματικά να προχωρήσω όταν είχαμε αρχικά την οδηγία του αμοιάντου στο κοινοβούλιο ήμουνα από εκείνους που είπαν πραγματικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί γιατί ξεκολουθούν να υπάρχουν εργαζόμενοι που πλήττονται από τον Αμιάντο και θέλω να ξέρω τι έγινε, πώς εξετάζεται το τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη, πώς εφαρμόζεται η τρέχουσα οδηγία για τον αμίαντο. ή μπορείτε να κάνετε και περίτερο έργο εδώ. Αυτά για να προφτάσετε και να απαντήσετε. σε ευχαριστώ. Η κυρία Γεσλοφέτσια. Και μετά θα υποβάλω και εγώ μια ερώτηση. Ε, ευχαριστώ. Η θέση του Διευθυντή, η όλη σας σταδιοδρομία, φανερώνουν ότι έχετε όλα τα παρέτα προσόντα για να αναλάβετε αυτήν την θέση. να σχολιάσω κάτι που έθιξε και η κυρία Ντελή. Είπε ότι σήμερα η αγορά εργασία επιβάλλει όλο και πιο αυξημένε απαιτήσει. Νέα επαγγέλματα, φόρτο εργασία από τη μια και από την άλλη παράταση του ορίου συνταξιδότηση. Αυτό σημαίνει ότι για τους πιο ηλικιωμένους οι δυσκολίες αυξάνονται. Από την πείρα σας λοιπόν θεωρείτε ότι ο οργανισμός σας μπορεί να στηρίξει τα κράτη-μέλη προκειμένου να θεσπίσουν τέτοια μέσα που να διευκολύνεται η πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες και μάλιστα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να παραμένει ποιοτική υγειονομική περίθαλψη ακόμη και να φτάσουμε στα 65, στα 67, στα 70, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι αποτελεσματικοί, επαγγελματικώς ενεργοί και να μην είναι εκτεθειμένοι στο εργασιακό άγχος. Πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα νέα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχετε πάρει το μολύβι σας και να έχετε σημειώσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Καταιγισμός. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Στην ε, προκατακτική σας ομιλία μιλήσατε και για τις δημογραφικές υποκλήσεις και το συσχετισμό τους με τα θέματα υγείας, ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει ώστε το 2012 να είναι το έτος της ενεργούς γύρανσης. Έχοντας λοιπόν κατά νου το στοιχείο αυτό εσείς πώς θα συμβάλλετε σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Και μια δεύτερη ερώτηση. Πώς θα καλύψετε τα του εργασιακού άγχους. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με του συντάκτε τη δική μα τη μελέτη, οι οποίοι μα είπαν ότι τελικά είναι πολύ λίγα τα στοιχεία που πραγματικά διαθέτουμε για το εργασιακό άγχο. Οι αναλύσει, τα, τα δεδομένα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τρόπο που συλλέγονται δεν είναι ακόμη επαρκή. Αυτή λοιπόν η ανησυχία απασχολεί όλο και περισσότερο μεν και Υπάρχει σοβαρό αντίκτυπο για το πώς λειτουργούν οι μισθωτοί εργαζόμενοι στις θέσει εργασίας τους. Προβλέπετε λοιπόν κάτι ιδιαίτερο για αυτόν τον τομέα. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με τη σειρά που θέλετε και με, όποια, με όποιο ενθουσιασμό εσεί κρίνετε κατάλληλο. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα με συμπληρώσετε αν κάτι ξεχάσω. Απλώς θα ακολουθήσω τη χρονική σειρά. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τα πρότυπα ή τέλο πάντων γενικότερα τον χρόνο εργασίας. Από νομοθετικής άποψης νομίζω ότι είναι αμφιλεγόμενο το όλο θέμα και η συγκεκριμένη οδηγία. Να σας πω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω κάνει εγώ συγκεκριμένα, για τις ώρες εργασίας και την επισφαλή εργασία, καθώς και τις δημογραφικές προκλήσεις. Αυτά τα θέματα κυρίως μας απασχόλησαν. Προφανώς η διάρκεια του χρόνου, ο χρόνος ακριβώς εργασίας είναι ένας παράγων που επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια. Στην εργασία όμως, ο χρόνος εργασίας πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για όλα τα ερωτήματα που ακούσαμε σήμερα. Μπορώ να πω ότι βάση για την ε, βελτίωση των ε, συνθήκων εργασίας στην Ευρώπη θα είναι να επιμείνουμε στην ε, πρόληψη, στο στάδιο της πρόληψης, να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την, ορθή, την σωστότερη προσέγγιση και να προάγουμε την ε, προστασία των εργαζομένων, να δημιουργηθεί μια κατάλληλη νοοτροπία. Εάν μιλάμε για χρόνο εργασία, εάν μιλάμε για ατυχήματα, εάν έχουμε τη σωστή νοοτροπία, τη σωστή προσέγγιση, όλα αυτά μπορούμε να τα διαχειριστούμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, όποιο κίνδυνο και αν ε, σκεφτούμε. Με ρωτάτε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του χρόνου εργασίας θα πρέπει να δω πληροφορίες και τις θα πρέπει να δούμε τις πληροφορίες και τις ορθές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται σε κράτη-μέλη. Έχω εργαστεί στην Αυστρία, την Γερμανία και την Ισπανία και γνωρίζω αρκετά καλά τα συστήματά τους και σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες επίσης έχω κάποιες γνώσεις και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ καλά πρότυπα για τον χρόνο εργασίας, και την κατανομή των, ε, του χρόνου εργασίας κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου. Ακόμα και σε σχέση με τις δημογραφικές αλλαγές θα πρέπει να αναλύσουμε και να διαδώσουμε τις καλές εμπειρίες και τις ε, χρήσιμες γνώσεις που διαθέτουμε. Και επίσης να δούμε τι παρεμβάσεις χρειάζονται σε επίπεδο επιχειρήσεων. Πάντως, το θέμα του χρόνου εργασίας είναι κάτι που νομίζω ότι και στο επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να απασχολήσει. Νομίζω ότι εδώ ο οργανισμός μας μπορεί να δώσει πολλέ χρήσιμε πληροφορίε. Επόμενη ερώτηση και παρακαλώ αν κάτι μου διαφύγει να μου το επισημάνετε έπειτα. Επόμενη ερώτηση ήταν αυτή για τον αμίαντο. Όταν διάβασα το τι κάνει τώρα ο Καναδάς για το θέμα αυτό, πραγματικά που αισθάνθηκα απογοήτευση. Διότι αυτό το έχουμε ξαναδεί στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι αρκετοί εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στον αμίαντο. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε είναι αυτής εξ αρχής να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον το ξέρουμε ότι μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε σε όλους τους τομείς και τους κλάδους. Ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό, πολλές χώρες το έχουν κάνει ήδη. Ο αμύαντος δεν μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα υλικό και αυτό είναι κάτι που πρέπει απλώς να φροντίσουμε να μαθευτεί. Πρέπει να συνεργαστούμε και με συνδικαλιστικές οργανώσεις και με ενώσεις εργοδοτών γιατί και αυτοί υποστηρίζουν ε, τέτοιες κινήσεις. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να διαδώσουμε τις, ε, τις ε, κατάλληλες πληροφορίες, έπειτα να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστα δεδομένα και τέλος να τονίσουμε το πόσο καλά παραδείγματα αντικατάστασης του αμύαντου έχουμε. Έπειτα για την Γερμανίδα βουλευτή και την ερώτησή της για τις νέες πρωτοβουλίες στη Γερμανία για την ποιότητα της εργασίας. Πρώτα απ' όλα, βάση εργασιών μας, είναι το τριμερές, ε, η τριμερής προσέγγιση, τρίπτυχο. Ε, εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε με συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών και ασφαλιστικές εταιρείες και μετά από κάποια χρόνια στη Γερμανία αυτό που πετύχαμε είναι να εμπλέξουμε στην όλη προσπάθεια και τις ίδιες τις εταιρείε, Να αναπτύξουμε από κοινού θηλυκές προς το χρήστη λύσεις. Από τις εταιρείε, ζητήσαμε να μάθουμε τι χρειάζονται. Η συνεργασία και η στήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ενώσεων εργοδοτών ήταν ένα από του παράγοντες που επέτρεψαν να πετύχουμε. Προσπαθούμε εδώ να έχουμε μια προσέγγιση όσο το δυνατόν σφαιρικότερη. Προσπαθούμε κάποια μηνύματα να είναι σαφή. Θέλουμε να υπάρχει μια νοοτροπία πρόληψη στι εταιρείε. Και η πείρα μου, ακόμα και με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, δείχνει ότι Βεβαίω θέλουν να έχουν ε, την σωστή νοοτροπία αντιμετώπιση του θέματος και εκείνοι, όμως χρειάζονται περισσότερη στήριξη, άρα πόρους, άρα και χρόνο. Αυτή νομίζω είναι οι παράγοντες που επέτρεψαν αυτή η πρωτοβουλία να είναι τόσο επιτυχής. Κάτι άλλο που σημείωσα είναι η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Επίσης, πώς τον γυράσκοντα πληθυσμό μπορούμε να τον ενθαρρύνουμε και να τον διευκολύνουμε ώστε να παραμείνει υγιής. Αυτό ήταν μέρος του έργου που θα αναλάβει στο παρελθόν. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι δημογραφικές αλλαγές δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι μεγαλύτερη ηλικία. Ήδη για τους νεότερους πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες. Οι νεότεροι πρέπει να κατανοήσουν τι σημαίνει υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε τις προσπάθειές μας, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ασχολούμαστε με τους νέους. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Επίσης, την εργασιακή ασφάλεια και υγεία γενικότερα πρέπει να τις προωθήσουμε, διότι κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου είναι σημαντικό να περιορίζονται κίνδυνοι και να προωθείται η υγεία. Λόγω χάρη στην πρωτοβουλία μας αξιοποιούμε διάφορα μέσα για την καλή διαχείριση ε, της εργασίας. Δηλαδή κοιτάζουμε πώς να επηρεάσουμε και τη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας αλλά και με μέτρα ισόρροπα που έχουν να κάνουν με, την, με τον ίδιο τον χώρο αυτό εργασίας. Νομίζω και οι δύο αυτές πτυχές είναι σημαντικές, διότι ξέρουμε ότι οι αριθμοί του του πληθυσμού αυξάνονται όλο και περισσότερο και αλλάζουν, ε, επιβράζονται πολύ τα πράγματα και από τι συμπεριφορέ της ατομικέ των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, ο οργανισμός μας ήδη μελετά το θέμα των ε, μεγαλύτερων σε ηλικία και των των εργαζομένων και θα πρέπει να σκεφτούμε κατάλληλα παραδείγματα για το πώς θα επηρεάσουμε τις εργασιακές συνθήκες, κυρίως για τους ε, μεγαλύτερους ηλικία εργαζομένους, όπως το άγχος, ε, το εργασιακό άγχος βλέπουμε ότι επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τους μεγαλύτερους από τους νεότερους και οι σωματικές τους ικανότητες είναι περιορισμένες. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να μάθουμε και μετά να προσαρμόσουμε τις εργασιακές συνθήκες σε αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν. Μια άλλη ερώτηση αφορούσε το 2012 ως έτος της ενεργούς γύρανσης. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις όπως η προσπάθεια ε, διάδοσης και ενημέρωσης, διάδοσης πληροφοριών και ενημέρωσης για θέματα των ε, γυρασκόντων εργαζομένων, των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και νομίζω ότι εδώ σημαντικό είναι παραδείγματα στρατηγικές ή πολιτικές που γνωρίζουμε από τα κράτη-μέλη να τις προβάλλουμε ως καλά παραδείγματα για να στηρίξουμε τους μεγαλύτερους ηλικία εργαζόμενους ή να επηρεάσουμε τις ε, ενώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών. Είναι και αυτό μια ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχω παρακολουθήσει με λεπτομέρεια όλες τις ε, δραστηριότητε, αλλά ξέρω ότι κάποιες ήδη ε, έχουν ξεκινήσει. Τώρα, το άγχος. Ένα θέμα πραγματικά πολύ σοβαρό και περίπλοκο. Θα γνωρίζετε ποια ήταν τα πορίσματα του κοινωνικού διαλόγου και τι έγινε με την υλοποίηση μέτρων για την καταπολέμηση του άγχους. Στη Γερμανία συγκεκριμένα υπάρχουν Υπάρχουν προβλήματα και παραμένει η ανάγκη βελτίωσης της κατανόησης των παραγόντων που επηρεάζουν στο χώρο εργασίας. Πρέπει να αναζητήσουμε εργαλεία και μέσα για να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση που επικρατεί σε ένα χώρο εργασία λόγω άγχου. Εδώ ο οργανισμό μα έχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνει. Μα περιμένει δουλειά γιατί είναι πολλά τα εργαλεία που υπάρχουν ήδη, αλλά δεν έχουμε αποτιμήσει τη λειτουργία του. Δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστα είναι για να τα προτείνουμε στη συνέχεια και στα κράτη-μέλη. Ίσως να μου θυμίζατε αν κάτι μου διέφυγε. Ναι. ναι για την αξιολόγηση του κινδύνου για τις ΜΜΕ. Ναι, αυτή η αξιολόγηση online ε, είναι κάτι που προετοιμάστηκε στις ε, κάτω χώρες. Είναι ένα μέσο λογισμικού που έχει σαν στόχο καταρχήν διάφορους κινδύνους και κατά δεύτερον διάφορους κλάδους και αυτό γίνεται με τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε οι ΜΜΕ εύκολα να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν αυτή την μέθοδο. Και η αξιολόγηση γίνεται σχετικά γλίγορα, είναι ευνόητη, έχει εξελιχθεί περαιτέρω στην υπηρεσία μας, έγινε ήδη μία δοκιμαστική προσπάθεια με συνεργασία εταιριών. Τα αποτελέσματα νομίζω ήταν μάλλον θετικά και είναι δυνατό να προσαρμοστεί αυτό στους διάφορους γλώσσες φυσικά και στη διαφορετική νομοθεσία από χώρα σε χώρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρχει πρόσβαση εκεί και να χρησιμοποιηθεί από ΜΜΕ. Πρέπει να γίνουν και άλλες δοκιμές ίσως, αλλά αυτό νομίζω ότι θα είναι ένα από τα μέσα που θα μπορούν να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σαν ένα πρότυπο να προσαρμόζεται μετά στις ανάγκες των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη από εκεί και πέρα θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για τις εταιρείε τους. Πρόεδρος, νομίζατε ότι τελειώσατε, αλλά έχουμε ένα συνάδελφο που ήρθε αργότερα και θέλει επίση να συμβάλλει στη συζήτηση. Θα τη ζήσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Άπτη. Εγώ ζητώ συγγνώμη και λυπάμαι που δεν μπορούσα να είμαι εδώ από την αρχή για λόγους ε, πέρα από τη θέλησή μου. Ε, να πω καταρχήν ότι χαίρομαι ιδιαίτερα να βλέπω μία γυναίκα υποψήφια για αυτό το τόσο σημαντικό πόστο. Να πω επίσης ότι όταν ήταν το συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Συνδικάτων στην Αθήνα, είχα περάσει από το περίπτερο του οργανισμού αυτού και είχα δει όλα όσα μέχρι στιγμής κάνουν. Οι απαντήσεις που άκουσα από τη στιγμή που ήρθα σε σχέση και με αυτά που είδα στο περίπτερο της Αθήνας αισθάνομαι ότι α, κουμπώνουν, ταιριάζουν, δένονται και θα δώσουν ένα πολύ καλύτερο μέλλον στον οργανισμό. Ε, μία πολύ μικρή ερώτηση, γιατί διάφορα άλλα πράγματα που είχα κατά νου ήδη τα αναφέρατε. Η Κομισιόν, προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της α, υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, χρησιμοποιεί διάφορες συμβουλευτικές επιτροπές, διάφορα σώματα. Ε, για παράδειγμα, αναφέρω το Advisory Committee of Health and Safety at Work ή το Senior Labor Inspectors Committee. Ε, η ερώτηση μου είναι πόσο αποτελεσματική θεωρείτε ότι είναι η δουλειά αυτών των επιτροπών, πόσο μπορεί να βελτιωθεί και τι θα είχατε να συμβουλεύσετε αυτές τις επιτροπές ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να μην είναι απλώς μία μελέτη κάνουμε μία μελέτη επειδή πρέπει να την κάνουμε και μένει στα χαρτιά. Αυτή η μελέτη να έχει σχέση ε, με, με, την, με την πράξη, με τον εργαζόμενο μέσα στη δουλειά του. Να μην μένει στα χαρτιά. Ευχαριστώ. I hope I understood you right. You... Λοιπόν, ε, αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε πώς βλέπω εγώ τη συνεργασία με αυτή εδώ την Επιτροπή. Ναι, αυτό που ρώτησα είναι πώς βλέπετε τη συνεργασία ε, με την Κομισιόν και με τις επιτροπές, τις συμβουλευτικές επιτροπές μελετών που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας στην εργασία. Uh, I Ελπίζω να σας κατάλαβα σωστά. Αυτό που χρειαζόμαστε γιατί αναφερθήκατε στην Κομισιόν και Συμβουλευτικές Επιτροπές, θα πρέπει να υπάρχει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα ανταλλαγή απόψεων. Και η Κομισιόν και όλες οι επιτροπές θα πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες, τι χρειάζεται στην εργασία τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ έχω συνηθίσει να εργάζομαι δίκτυα και ξέρω ότι η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Υπήρξε λοιπόν τακτική επικοινωνία και σαφής ανταλλαγή πληροφοριών και πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες. Μόνο αν ξέρουμε τις ανάγκες μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια. Αυτό είναι σημαντικό νομίζω. Αυτά προς το παρόν. Αυτό ρωτήσατε αν δεν κάνω λάθος και δεν έχω να σας απαντήσω τίποτα άλλο. Can you, uh, conclude? Θέλετε να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Ναι, φυσικά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μου δώσετε τη δυνατότητα να είμαι εδώ και να ακούσω πώς λειτουργεί αυτή η Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τακτική ανταλλαγή απόψεων άκουσα ότι είναι δύσκολο να ακολουθήσω τον προκάτοχό μου, το ξέρω βέβαια, ξέρω ότι το γνωρίζω τον κύριο Τάκαλα εδώ και πολύ καιρό, νομίζω ότι έχουμε παρόμοια προσέγγιση στο θέμα της εργασιακής ε, ασφάλειας και υγείας, αλλά πολλά αλλάζουν βέβαια στον χώρο της εργασίας που αλλάζει σήμερα. Χρειάζονται νέα μέσα για να αντιμετωπιστούν τα νέα προβλήματα θα κάνω ό,τι μπορώ και θα προσπαθήσω να έχω πολύ καλή και διαφανή επικοινωνία και με εσείς και με άλλες επιτροπές. Γιατί θεωρώ ότι προστιθέμενη αξία της συνεργασίας στο δικό σας επίπεδο είναι να υπάρχουν πληροφορίες από διαφορετικές σκοπιές. Αυτό είναι ακριβώς η προστιθέμενη αξία πάνω σε αυτή θα πρέπει να βασιστούμε και να εργαστούμε. Και η υπηρεσία μας εργάζεται προς την αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και να έχουμε τακτή επαφή μαζί σας για να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια κάστοτε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ελπίζω να ξαναειδωθούμε συχνά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι θα ξενιδωθούμε. Αν κατάλαβα θα αναλάβετε το καθήκοντά στις 15 Σεπτεμβρίου. Και μέχρι τότε θα είσαστε πλήρως έτοιμοι φαντάζομαι για να λάβετε τις ευθύνες σας. Μια που κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε για μια μεταβατική περίοδο, ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τάκαλα για να μας πει τι έγινε. Ε, ποιες είναι οι εμπειρίες του με το την υπηρεσία του Μπιλμπάου. Ξέρω θα παρέμβετε στο σημείο 23 ημέρε τη διάταξη, αλλά δεν θα είμαι πλέον παρούσα και θα ήθελα να σα ακούσω τώρα, αν έχετε να πείτε δύο λόγια. Ωραία. Θα πείτε ότι έχετε να πείτε αργότερα που θα λείπω εγώ, αλλά θα μου πούν οι συνάδελφοι τι θα έχετε πει. Euh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας κυρία μου και σας ευχόμεθα κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο της διάταξης και περνάμε στο επόμενο σημείο. Σημείο 20. Θα ήθελα να δώσω το λόγο εδώ στον Θοδωρικ Ταρντέν για την παρουσίαση των τροπολογιών για το σχέδιο εκθεθεί στο πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα την Καταπολέμηση Φτώχεια και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Για το θέμα αυτό έλαβε 396 τροπολογίες. Ε, τουλάχιστον αυτό αποδεικνύει μεγάλη επιτυχία ενδιαφέροντος. Τώρα ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσμα δεν ξέρω. Ευχαριστώ, Madame Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως είπατε είναι πάρα πολλές οι από όλες τις πολιτικές ομάδες. Η δική μου η ομάδα των σοσιαλιστών των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Νομίζω ότι είναι γνωστή για το ότι δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις απόψεις όλων των συναδέλφων. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε από τώρα ήσυχοι γι' αυτό. Και για το σχέδιο έκθεσης να πω ότι δεν μπορέσαμε να τα καλύψουμε όλα σε αυτό το σχέδιο. Ιδίω λόγω του πόσο ευρεία είναι η προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ το περιθώριο που έχουμε είναι πολύ στενό. Εγώ ο ίδιος από τροπολογίες μόνο έχω υπογράψει 70 τέτοιες. Είναι πάρα πολλές όλες από τους υπόλοιπους συναδέλφους. 396. Καταλαβαίνουμε παρόλα αυτά ότι οι περισσότερες εμπλουτίζουν ε, την τελική έκθεση και μάλιστα συγκλίνουν σε πολλά σημεία. Οπότε θα έχουμε έτσι πολλές καλές δυνατότητες να πετύχουμε συμβαστικές λύσεις για πολλά θέματα, όπως το πώς θα καλύπτονται οι συμβαλόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι και όσοι βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας. Επίσης, η ενεργός συμμετοχή και σχετικές ρήτρες, η δημιουργία πλατφόρμας με δείκτες ένα κράτος μέλος, θέματα που επανέρχονται και επαναλαμβάνονται σε πολλές τροπολογίες. Ένα θέμα που επίσης τυχαίνει να είναι επίκαιρο. Επισητιστική βοήθεια για τους ε, μειονεκτούντες. Παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων λόγω συνθήκων φτώχειας και επίσης το καλάθι των βασικών αναγκών. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια θέματα, κάποιες μέρημνες που διέπουν όλες τις ομάδες, τις, στις προτεραιότητές τους. Θα φροντίσουμε λοιπόν η έκθεση αυτή παρόλα αυτά να παραμείνει κατανοητή, εύληπτη. Τροπολογίες που εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συνδυαστούν σε τέτοιες συμβαστικές λύσεις ώστε να διαρθρωθούν καλύτερα οι ιδέες που προτείνονται αλλά δεν θα είναι και τόσο εύκολο, διότι κάποια θεματάκια θα είναι κάπως πιο δυσχερή. Κανένας δεν θα εκπλαγεί που η νομική ασφάλεια της Επιτροπής για την υλοποίηση της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας λόγω χάρη θα είναι ένα από αυτά. Ή η αρμοδιότητα της Ένωσης, όταν μιλάμε για το ελάχιστο εισόδημα, το τι μισθό υπάρχει μεταξύ του όρου μισθός, ε, ελάχιστο εισόδημα. Πρέπει εδώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους όρους που και λόγω των μεταφράσεων αλλάζουν. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σίγουρα επανειλημμένος. Επίσης η απεμπλοκή της ε, οδηγίας, οριζόντιας οδηγίας και το τι επιπτώσεις θα έχει η δέσμη μέτρων ε, για την οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν, ελπίζω, να προχωρήσουμε στον προβληματισμό μας και νομίζω ότι όταν δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τα φαινόμενα φτώχειας και να προτείνουμε καινοτόμε και φιλόδοξες λύσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερος λοιπόν που και οι Υπουργοί που χθε μόλι ε, μίλησαν για το θέμα αυτό στο σώμα μας, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους. Εδώ, Πρόεδρε, η γενική μας άποψη για την τροπολογία. Λείπουν κάποιοι από του συναδέλφου που τροπολογίε. Παρ' όλα αυτά ας ανοίξουμε την συζήτηση. Η κυρία Λίν, μετά η κυρία Ντελή, η κυρία Λίν. Ναι, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας και φυσικά και για το γεγονό ότι χρειάστηκε να διαβάσει 496 τροπολογίε. Εγώ τις ε, διάβασα ε, και πρέπει να σας πω ότι χρειάστηκα 3,5 ώρες για να διαβάσω και τι 396, Επομένω, πρόκειται για αρκετή δουλειά. Έχω εντοπίσει κάποιους τομείς οι οποίοι μπορεί να μας δημιουργήσουν ε, πρόβλημα. Το διαθέσιμο εισόδημα είναι σημαντικό. Χαίρομαι που κάναμε διαχωρισμό μεταξύ ελάχιστου εισοδήματος και ελάχιστου μισθού διότι είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί την Επιτροπή και ε, υπάρχουν και προβλήματα με τις μεταφράσεις επ' αυτού. Όταν μιλάμε για ελάχιστο εισόδημα, μιλάμε απλώς για τα κοινωνικά επιδόματα, ε, επιδόματα από το κράτος μέλος και όχι από τον εργοδότη ως ελάχιστο μισθό. Η ομάδα μου βεβαίως δεν θα ήθελε να υπάρχει νομοθεσία για το ελάχιστο εισόδημα, εγώ το υποστηρίζω. Θεωρώ ότι το ελάχιστο εισόδημα για όλα τα κράτη-μέλη είναι εξαιρετική ιδέα και κάθε κράτος μέλος που δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να έχει ελάχιστο εισόδημα στο κράτος του θα πρέπει να το κάνει. Αλλά αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει από κοινού με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν νομίζω ότι χρειάζεται νομοθεσία απαραίτητο γι' αυτό το λόγο για την 359, την 366, την 387 ε, και την 368 έχω κάποια προβλήματα, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Επίσης να σας πω ότι θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ των πολιτικών ομάδων αλλά και εντός των πολιτικών ομάδων. Οι 381 και οι 386 που ζητούν ε, μια οδηγία πλαίσιο για τις ε, ε, υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος και κοινή ωφελία είναι κάτι το οποίο μας αποσχολεί. Η ομάδα μου δεν είναι υπέρ μιας οδηγίας για τις υπηρεσίες κοινή ωφελίας θα τις καταψηφίσουμε αντιστοίχως και για την 320 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη εμείς πάντα ήμασταν της έποψης ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να γίνεται επί εθελουσίας βάσεως και δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάτι νομοθετικά για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πέραν όμως αυτών των σημείων που νομίζω ότι πολλά μέλη στην Επιτροπή έχουν αντίθετη άποψη. Ε, πολλές από τις τροπολογίες είναι πολύ καλές και προσθέτουν και κάποια στοιχεία στην έκθεσή σας. Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να δούμε περισσότερες τροπολογίες εκ των προτέρων, διότι αν συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τόσους πολλές τροπολογίες από, σε κάθε έκθεση, ε, θα υπάρχει πρόβλημα και νομίζω ότι το πρόβλημα δημιουργείται και από τον τρόπο που κατατίθεται πλέον η τροπολογία. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιο ε, παρόν και να προσθέσει την υπογραφή του. Μπορεί κάποιο να καταθέσει πλέον τροπολογία χωρί να είναι παρόν για να την ε, υπερασπιστεί ή να χρειαστεί και να την υπογράψει. Ελπίζω να μην έχουμε τόσες πολλές τροπολογίες ε, στα επόμενα ζητήματα, γιατί όσοι μας ασχολούνται με οδηγίες και εκθέσεις ε, ή και γνωμοδοτήσεις ε, θα έχουν πολύ προβλήματα να καταλήξουν σε συμβιβαστικέ προτάσεις από κοινού. Επειδή ακριβώς θα έχουμε δε και το καλοκαιρινό διάλειμμα, για μας θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Υπάρχει βεβαίω πάντα τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα. Ξέρω ότι το θέμα πρέπει να είναι έτοιμο για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας για τις τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν ελεύθερα επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί μου ε, και θα προσπαθήσουμε να ε, κάνουμε κάτι από κοινού ώστε να έχουμε μια καλή έκθεση στο αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που ήθελα να αναφέρω εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Κύριε euh, euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε. Έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, νομίζω, και πολλές κοινέ τροπολογίες. Είναι πολύ καλό αυτό. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του κατεπήγοντος. Ε, μέσα στο, στην έκθεση αυτή επιμένουμε στην διατήρηση του επιστημικού ε, προγράμματος γιατί οι περικοπές της Κομισιόν είναι απαράδεκτα. Πρέπει να εγγυθούμε στην επιστημική τράπεζα σήμερα <clears throat> τις επιδοτήσεις που έχει. Αλλιώς δεν θα ξέρει αύριο πώς θα διαθρέψει χιλιάδες χιλιάδων ατόμων αυτή η πολιτική της καταπολέμησης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού περνάει και το λέω το σωστά στην έκθεσή σας από νέα ατζέντα κοινωνικών θεμάτων και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να τονίσουμε μόνο το, την απασχόληση γιατί σήμερα μιλάμε πολύ για τους φτωχούς εργαζόμενους και το λέει η έκθεσή σας. Πρέπει να επιθυμίσουμε τι είναι η ελληνική. Η ελληνική είναι προς εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από τους συμπολίτε μας. Ε, λέγεται ότι θα είναι 20 εκατομμύρια αυτά τα έτομα θέλει να μειώσει η Κομισιόν σε 20 εκατομμύρια μάλλον. Μου φαίνεται πολύ φιλόδοξο αυτό το σχέδιο προσωπικά. Αλλά αν έχουμε την τόλμη και αυτό το συμφωνώ μαζί σας κυρία Κλήρ, να έχουμε τα μέσα για να το πετύχουμε, ιδίω ενός νομοθετικού πλαισίου για το σύστημα ελαχίστου εισοδήματος, ούτω ώστε ο κάθε πολίτης να έχει ένα βασικό εισόδημα για να μπορεί από εκεί και πέρα να αναπνεύσει και να βγει από την κατάσταση φτώχειας να έχει δηλαδή κατάλληλο εισόδημα για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του ε, τροφή, νερό, πρόσβαση στις ε, δημόσιες μεταφορές κλπ. Αυτό θα ήταν μεγάλο βήμα για την κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σπουλό. Και εκεί μετά ο κύριο Κοσλόφσκι. Θα είναι πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Είναι τεχνική μορφή η παρεμβασή του. Είμαι σίγουρο ότι θα βρούμε συμβασμού με τον κύριο Τερντέν. συμβαστικέ λύσει μια που η, η έκθεση του είναι υψηλωτά της ε, ποιότητα. Εγώ υπέβαλα δύο τροπολογίε για την 101 και 102 κάπω εκ των υστέρων. Ζήτησα να τοποθεθούν στο 19α και 19β αν είναι δυνατόν προς το τέλος δηλαδή. Αυτό είναι ένα αίτημα που θέλω να επαναλάβω προφορικά. Ευχαριστώ κύριε Κοσλόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για το έργο του. Και παρεμπιπτόντως να ευχαριστήσω και την σκιώδη εισηγήτρια που ζητά συγγνώμη για τη σημερινή της απουσία. Μιλώ λοιπόν και εκ μέρους της. Ε, έκανε σημαντική δουλειά ε, στην κατάθεση των τροπολογιών και θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία, πολύ σύντομα. Σημείο 9 της έκθεσης προτείνω να υπάρχει αναφορά στις εγγυήσεις για τους εργαζομένους εγγυήσεις για τα δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να απολεμβάνουν ε, σε κοινωνικές εισφορές. δεν είναι πάντα οι ίδιες λύσεις οι κατάλληλες για τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ επίσης την προσοχή και στην παράγραφο 18 της έκθεσης για την έκθεση πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα. Θεωρώ ότι το θέμα της ένδυας είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και επομένως θα πρέπει να έχουμε μία ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Το θέμα της παιδικής φτώχειας τώρα. Ένα φρικτό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει και μακροπρόθεσμα πολύ δραματικές συνέπειες. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι πολύ συχνά η παιδική φτώχεια ε, έχει άμεση σχέση και με τη φτώχεια της ίδιας της οικογένειας. Επομένως θα πρέπει να βρούμε κανόνες που να στηρίζουν όλη την οικογένεια. Κάποιες από τις τροπολογίες μου οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση η ιδίω στην αιτιολογική σκέψη L και η τροπολογία που κατέθεσε στην παράγραφο 17. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Η συνάδελφο Ελίζα να αναφέρθηκε στην κοινωνική και περιφερειακή ευθύνη των επιχειρήσεων. Ένα θέμα που συχνά έχουμε δείξει στην Επιτροπή αυτή και πάνω στο οποίο ξέρω ότι τάση δεν είναι εκείνη που θα ήθελα. Θα ήθελα απλώς να πω όμως ότι ακόμα και από την πλευρά των επιχειρήσεων δεν συμμερίζονται όλοι την προσέγγιση της Business Europe. Και σήμερα ακριβώ είχα μια συνάντηση με προσώπους των ειδικευμένων λογιστών που αναφέρονται κατά του υποχρεωτικού χαρακτήρα αυτών των διατάξεων. Δεν ξέρω λοιπόν πάντα θα πρέπει να μιλάμε για πολυεθνικές και τις εκπροσωπήσεις τους στα κράτη-μέλη. Τέλος πάντων αυτό είναι μια συζήτηση που ξέρω ότι θα συνεχίσει να μας ανησυχεί εδώ στην Επιτροπή μας. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διάφορους περιβαίνοντες που επέσαν την προσοχή μου εκ νέου σε διάφορα σημεία που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και ομολογώ ότι θα είμαι πολύ προσεκτικός ε, όσον αφορά το συμβιβασμό και όσον αφορά την ανάλυση εις βάθος των διαφορών τροπολογιών. Και θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω για τις ανησυχίες του, αλλά και για τη διαθεσιμότητά τους για τον φάκελο αυτό. Λόγω των θερινών διακοπών, ίσως τα χρονικά όρια θα είναι πολύ στενά και η πρόταση της κυρίας Λίν να προσπαθήσουμε ήδη να βελτιώσουμε την επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλή η πρόταση. Δεν θέλω να επιθέσω τώρα στα διάφορα θέματα που εθίγησαν, που είναι συνενετικά εύκολα ή κάπως πιο δύσκολα ίσως, αλλά αναμενόμενο ήταν. Και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω τέλη Αυγούστου να συναντηθούμε με συμβαστικές προτάσεις για να εργαστούμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, Ευχαριστούμε. Άρα, με να σας ευχόμαστε καλό κουράγιο για την εξέβρεση συμβαστικών προτάσεων. Τι θα κάνουμε τώρα. Όλα μαζί. Όλες μας θα τις δούμε και πρέπει να έχουν εγκριθεί στις 8 Σεπτεμβρίου. Οπότε στην προηγούμενη συνεδρία που αναφέρατε πρέπει να έχουν ε, υποβληθεί τροπολογίες και θα ψηφίσουμε την έκθεσή σας στην δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Σημείο 22 τώρα της ημερήσιας διάταξης, νομίζω ο κύριος Έλμερ. Όχι, με συγχωρείτε, 21. Ο κύριος Έλμερ αντικαθιστά τον κύριο Κάμπλνοχ για την εξέταση του σχεδίου έκθεση για την εφαρμογή τη οδηγία 2536 σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Κυρία Έλμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε και εσείς και οι συνάδελφοι εκ μέρου του κυρίου Κάμπνο, ο οποίος έπρεπε να βρίσκεται στην ε, χώρα του σήμερα. Μου ζήτησε λοιπόν να σας παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Εδώ Μα απασχολεί η εφαρμογή τη οδηγία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Οδηγία που αφορά εξίσου την Επιτροπή εσωτερική αγορά. Εμείς όμως ετοιμάζουμε μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό και πρέπει να πω ότι δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα με την τωρινή εκδοχή της έκθεσης εκείνη την Επιτροπή. Πάντως ο κύριος ε, Κάμπνοχ έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις ε, γιατί πιστεύει κατά πρώτον ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εργαζομένων είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίση, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει να διευκολύνει την διασυνοριακή ε, κινητικότητα ώστε να διευκολυνθεί η εσωτερική αγορά και η πρόθεση τη ανάπτυξη και τη οικονομική αύξηση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζει την ανάγκη εξυγχρονισμού τη επικαιροποίηση μάλλον οδηγία 2005-36 ΕΚ, την προηγούμενη δηλαδή οδηγία. Είναι πεπισμένο ότι ο αριθμός των ε, ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων πρέπει να μειωθούν, ώστε να υπάρξει αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και σε νέους επαγγελματικούς κλάδους. Διεύρυνση λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς, στους καινοτόμους και την βιομηχανία τις καινοτόμες, τις τεχνολογίες και την, ε, τις σχετικές βιομηχανίες. Επίσης θα πρέπει το λεγόμενο IMI να προωθηθεί ώστε να υπάρχει ένα κεντρικό ε, διαλογικό πληροφορικό, εργαλείο πληροφορικής που να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό οι αρχές και το κοινό καθώς και εργαζόμενοι παρόλο ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων. Χρειάζονται ε, κανόνε αυτόματη αναγνώριση σε κάποιου τομεί, όπω του τεχνίτε ή σε κάποιου βιομηχανικού κλάδου και θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει την ε, καταγραφή και την έγκριση των επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένου κλάδου, χάνοντα τα κάτι μέλη να το αποδεχτούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα υποχρεωτικό ε, μητρό το οποίο να υλοποιείται για όσους η επαγγελματική άδειά τους έχει ανακληθεί από κάποιο κάτω μέλος. Και για τις αρχές των κατομελών θα πρέπει εδώ να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες. Ε, προσωπική μου παρατήρηση εδώ, ο το Ηνωμένο Βασίλειο ανέλαβε αμέσω δράση αναλόγω σε ένα σχετικό τομέα όταν ένα γιατρό που εξασκούσε το επάγγελμά του κατά τρόπο αθέμητο συνελήφθη να το κάνει αυτό στη Γερμανία. Ε, η άδειά του ανακλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίση θα πρέπει να υπάρχουν και γλωσσικέ απαιτήσει ε, και να υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία για τι ικανότητε ε, γλωσσικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και αυτό μπορεί να το απαιτεί ο εργοδότη μετά από ραντεβού από κανονισμένη συνάντηση. Θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κόστου σε όλα τα επίπεδα, ιδίω αυτό που καταβάλουν οι ίδιοι επαγγελματίε. Νομίζω ότι ούτε η έκθεση ω έχει ε, και όπω έχει διαμορφωθεί στην Επιτροπή Ιστορικής Αγορά, ούτε. Είμαι πολύ αισιόδοξο εδώ. Ούτε οι προτάσει λοιπόν του κ. Κάμπνοχ θα προκαλέσουν ιδιαίτερε διαφωνίε. Είμαι έτοιμο να ακούσω τι απόψει των μελών τη Επιτροπή. Κυρία έτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα βασικά προνόμια που απορρέουν από την ολοκλήρωση. Για να βγούμε από την οικονομική και χρηματοπιστωτική χρήση πρέπει να υποστηρίξουμε την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και γρήγορα στις ανάγκες των αγορών εργασίας των κρατών μελών. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι εδώ και πολύ καιρό ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το στοιχείο της ελεύθερης μετακίνησης, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά προσκόμματα ε, λόγω και της μεγάλης ποικιλομορφίας της ε, νομοθεσίας ε, στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό μόλις 1-2% και κάτι ε, ε, των πολιτών επωφελείται αυτής της δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε δραστηριότητες υπέρ της ε, κινητικότητας διαμεθοριακά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης που διατύπωσε μια εξαιρετική γνωμοδότηση που συντάχθη υπέρ της ε, διαμεθοριακής κινητικότητας, κάτι το οποίο θεωρώ πολύ θετικό βάσει και της πείρας που έχουμε από την εφαρμογή της, ε, επαγγελ... της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, θεωρούμε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απλούστευση των διαδικασιών, ε, σε πιο αυτόματο τρόπο αναγνώρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και όπου υπάρχει προσαρμογή στους νομοθετικούς κανόνες ε, στην σύγχρονη εποχή. Εξ του ΕΛΚ επικεντρώθηκα στα εξής ενίσχυση της ε, διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, διότι όπως λέει και ο ίδιος ο συντάκτης της νομοδότησης, θα πρέπει να υπάρχει απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του συστήματος για την εσωτερική αγορά, του EMI. Όπου υπάρχουν δυσκολίες, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ε, δυνατότητες συνδρομής των κρατών μελών. Είναι θεμελιώδη σημασία να επαληθεύουμε και να επικαιροποιούμε τι ελάχιστε απαιτήσει για την κατάρτιση κάποιων επαγγελματικών κατηγοριών. Όπω για παράδειγμα, ε, ιατρικά επαγγέλματα, νοσοκόμιο, οδοντοτεχνικοί διότι ε, οι απαιτήσει που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από τη δεκαετία του 70 και του 80. Θα πρέπει επίση να επικαιροποιήσουμε και τον κατάλογο των διπλωμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να διασφαλίσουμε ε, όσο το δυνατόν περισσότερη αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχει και πρόβλημα στην ε, ερμηνεία του άρθρου 11 ε, του επίπεδου των δεξιοτήτων και μπορεί να χρειάζονται και παρεκκλήσεις, να σκεφτούμε πιθανές παρεκκλήσεις για το άρθρο 11, ώστε να είναι πιο σαφές, ε, ε, πιο σαφές και πιο κατανοητό. Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί επίσης και τον κατάλογο των ρυθμισμένων επαγγελμάτων, όπου μπορούμε να έχουμε αυτόματη αναγνώριση των προσόντων. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε ακόμα μια φορά την ε, ιδέα μιας κοινή πλατφόρμας να διευκολύνουμε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Εξ όσων γνωρίζω, από τότε που ετέθησε ισχύ η οδηγία δεν υπάρχει καμία πλατφόρμα αυτή τη μορφή. γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιήσουμε την ε, νομοθεσία εν ισχύ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, προσβλέπω στη συνεργασία με το συντάκτη τη νομοδότησης και τους κοιόδης συντάκτες. Ευχαριστούμε κυρία Στάινμπροκ και μετά κυρία Τουρούνεν. το στοιχείο της ολοκλήρωσης στην αγορά εργασίας ε, έχει ως αναπόσπαστο τμήμα το την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πολλές από τις χώρες μέλη δεν έχουν ακόμα μεταφέρει την οδηγία και υπάρχουν προβλήματα με τους ε, τίτλους και τα διπλώματά τους. Όσον αφορά τώρα τη γνωμοδότηση, είναι μια πολύ καλή αρχή. Η συνάδελφος προηγουμένως ε, αναφέρθηκε σε κάποια σημεία με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Κατ' εμέ θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές ε, και η ομάδα των σοσιαλιστών θα καταθέσει και κάποιες τροπολογίες κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων όταν συζητάμε τα θέματα της απλούστευσης και εφαρμογής των διαδικασιών. Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο γρήγορη, πιο διάφανη αναγνώριση ε, όλων των επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα που ε, είναι νομικώς ρυθμισμένα. Η πλειονότητα των προβλημάτων βεβαίως προκύπτει από τα επαγγέλματα που δεν έχουν ε, ρύθμιση σε νομοθετικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα εθνικό σημείο επαφής για συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών, για διαβίβαση των πληροφοριών προς τους πολίτες και θεωρούμε ότι είναι ένα απαραίτητο βήμα. Εξυγχρονισμός της οδηγίας, ο οποίος θα πρέπει να μας ε, επιτρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ε, κάποιες πρωτοβουλίε οι οποίες υπάρχουν ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η διαδικασία της ε, Μπολόνια για, την, ε, για τις επαγγελματικές δεξιότητες στην Ευρώπη και υπάρχει και το θέμα της επίσημης αλλά και της άτυπης κατάρτισης. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και το θέμα της διαβίου μάθησης και κατάρτισης και ολοκληρώνοντας να πω ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανέναν έρμεο τις μοίρας τους, ακόμα και αυτοί που δεν αναγνωρίζονται τα προσόντα τους ή αναγνωρίζεται μόνο τμήμα των προσόντων τους, δεν θα πρέπει ε, να λησμονούνται. Θα πρέπει να ε, βρούμε ένα τρόπο να αντιμετωπίσουμε το κενό που διαπιστώνουμε στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε, η κυρία Τούρνεν. Καταρχάς ένα γενικό σχόλιο. Ως μέλος ε, της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ ε, ασχολούμαστε και εκεί με το θέμα αυτό. Η κατάσταση έχει ως εξή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έγγραφο εργασίας ε, του της που είναι καλό κατά την άποψή μου και έχει τύχει και μεγάλη υποστήριξη στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, αλλά είναι σαφές ότι το θέμα αυτό έχει και μια πολύ ισχυρή διάσταση απασχόλησης. Επομένως είναι λογικό να συμμετέχει ε, έντονα η Επιτροπή Απασχόλησης, ίσως και περισσότερο από τη συζήτηση που κάνουμε από αυτή τη στιγμή, ίσως να κάνουμε και κάποια συζήτηση κοινή με την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι δυνατό, αλλά νομίζω ότι είναι κοινό το ενδιαφέρον και των δύο επιτροπών μας. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία και θα καταθέσω και σχετικές τροπολογίες. Ε, παράγραφος 2. Υποστηρίζουμε πλήρω ε, τα όσα λέει παράγραφο 2, αποτελεσματική λειτουργία τη αγορά εργασία, ε, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κ.ο.κ. αλλά θα θέλαμε να προσθέσουμε και ότι υπάρχει ανάγκη για ε, την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ των σημείων αυτών και την ανάγκη να σκεφτούμε τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν με επαγγελματικού κανόνε που αιτιολογούνται λόγω δημοσίου συμφέροντος, όπω για παράδειγμα περιβαλλοντική προστασία, η προστασία και η ασφάλεια και η υγεία και όλα τα ζητήματα λοιπόν που μας αποσχολούν συνεχώς αυτό το αιώνιο δίλημα της ισορροπίας. Δεύτερον, ένα θέμα για την ε, κατάρτιση, την επιπλέον επιμόρφωση και την αναγνώριση της ε, κατάρτισης που γίνεται σε άλλες χώρες ε, μέλη και κάτι που περιλαμβάνεται στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επαγγελματικό στοιχείο, αυτό το professional cut, ε, θεωρούμε ότι είναι το νέο, η επαγγελματική κάρτα, συγγνώμη, το νέο ε, σημαντικό στοιχείο θα πρέπει αυτή η κάρτα ε, να έχει τη δέουσα αξία, να αξίζει κάτι και να υπάρχει ένα σύστημα που θα την υποστηρίζει. Δάλλος είναι άχρηστη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν θα θέλαμε να προσθεθούν τα στοιχεία αυτά στην ε, γνωμοδότηση. Βεβαίως αποτελεί καλό εφαλτήριο γνωμοδότηση και όπως είπατε και εσείς κύριε Χέλμ δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν και μεγάλες διχογνωμίες επί του θέματος. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν επιπλέον σχόλια, να δώσω το λόγο στον κύριο Χέλμ εξ ονόματος του συντάκτη της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους για την πολύ σημαντική συνεισφορά τους, ε, την οποία φυσικώς θα διαβιβάσω στον ε, κύριο Κάμπρινορχ, ο οποίος ε, θα δώσει και τη δέουσα προσοχή στα θέματα αυτά. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να περάσουμε Τώρα στην κατάθεση ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, συγγνώμη, 23 Αυγούστου το μεσημέρι, θα συζητηθεί την 1η Σεπτεμβρίου και έγκριση στις 19 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, επομένως, πολλή δουλειά και σε αυτό το θέμα για το καλοκαίρι. Τώρα, επειδή είμαστε πολύ προχωρημένοι στην ημερήσια διάταξη, αλλά ο κύριος David Michaels είναι ήδη εδώ, θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ντέιβιτ Μάικολς, ο οποίος είναι υφυπουργός εργασίας των ΗΠΑ, αρμόδιος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ε, είχε προσκληθεί στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσει τις πολιτικές ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της στρατηγικής 2007-2012 για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο της εργασίας, που συντάσσεται όπως ακούσαμε ε, από την κυρία Καρή Μαντελή. Θα σας δώσω το λόγο για περίπου 10 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με προσκεκλημένοι. Είναι τιμή για μένα και να σας απευθύνω το λόγο σήμερα. Χαίρομαι που βρίσκομαι στις Βρυξέλλε, που είναι διεθνής πόλη με μεγάλη ιστορία και είναι και κέντρο σεβασμού ε, για την επίλυση των προβλημάτων. Σας στέλνω χαιρετίσματα από την Υπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών ε, στα θέματα εργασία, τη Χίλντα Σόλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνει τη δυνατότητα να σας μιλήσω εδώ σήμερα. Θα σας μιλήσω για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο της εργασίας στις Ηνωμένε Πολιτείε και το πώς προσβλέπουμε στην ανάπτυξη μέσω συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι επιδημιολόγος. Έχω αφιερώσει το έργο μου στον εντοπισμό κινδύνων στον χώρο της εργασίας που μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους. Τώρα πλέον είμαι υπεύθυνο στο ε, Γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συνεργαστώ με τους Ευρωπαίους εταίρους μου. Φέτος εορτάζουμε την 40η επέτειο του οργανισμού μου. Πριν από 40 χρόνια το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ε, πέρασε το νόμο για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο της εργασίας και δημιούργησε ένα νέο βασικό δικαίωμα για τους εργαζομένους, το δικαίωμα σε ένα ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας. Σήμερα η χώρη εργασία στην Αμερική είναι πολύ πιο ασφαλής από ότι πριν από 40 χρόνια. Πριν από τον Όσα, περίπου 38 εργαζόμενοι την ημέρα σκοτώνονταν επί το έργο, ενώ σήμερα ε, με διπλάσιο εργατικό δυναμικό ο μέσο όρο είναι περίπου 12. Δυστυχώς όμως έχουμε επιτύχει παρά το πρόοδο, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μα. Πάνω από 4.500 εργαζόμενοι σκοτώνονται στο χώρο της εργασίας ε, κάθε χρόνο και κάθε χρόνο έχουμε αμέτρου τους ανθρώπους οι οποίοι τραυματίζονται, έχουν ε, εγκάφματα, ε, μελανόματα, ε, σπασμένο στά και ακροτηριασμούς. Και επομένω θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την κατάσταση και τα ατυχήματα στο χώρο της εργασίας. Αυτά όμως δεν είναι παρά μόνο στατιστικά στοιχεία. Ε, υπάρχουν και το κοινωνικό κόστος ε, που σχετίζεται με τους τραυματισμούς και τις ασθένειες στον χώρο της εργασίας και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, τα στατιστικά στοιχεία δεν πάβουν να είναι άνθρωποι που πάσχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε αντιμετωπίζουν πολλέ προκλήσει για την πρόληψη των ασθενειών και είμαστε εκτεθειμένοι καθημερινώ και σε πολυάριθμου χημικού κινδύνου. Εμφανίζονται και νέοι άγνωστοι κίνδυνοι. Ε, και το εργατικό δυναμικό γυράσκει. Ε, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο προσωρινούς, ε, προσωρινά απασχολούμενους ε, που είναι ανεκπαίδευτοι σε θέματα ασφάλειας και υπάρχουν και εργαζόμενοι ε, που έχουν ε, προβλήματα γλώσσας, γεγονός που αποτελεί επιπλέον εμπόδιο για την ασφάλεια και την υγεία τους. Η τελευταία πρόκληση είναι πολύ σημαντική για μας και στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα ε, προσεγγίσουμε αυτούς τους εργαζόμενους ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προστατεύονται. Μια άλλη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι και οι μικρές, ε, μικρές επιχειρήσεις ε, προστατεύουν αντιστοίχω τους εργαζομένους τους. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν υψηλότεροι κίνδυνοι, οι ε, ιδιοκτήτε μικρών επιχειρήσεων πολλέ φορέ δεν έχουν ε, πόρου για να καταρτήσουν ε, καταλήλω του εργαζομένου του και να διαχειριστούν του κινδύνου. Με τόσο λοιπόν πολλέ κοινέ προκλήσει, είναι λογικό να συνεργαστούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ λύσει. Το 1995 υπεγράφει μια νέα διατλαντική ατζέντα για να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά θέματα και από τότε υπάρχει μια ομάδα εργασίας για την απασχόληση και τα θέματα της εργασίας. Έχουμε οργανώσει συνεδριάσεις, εργαστήρια, διασκέψεις και ανταλλάσσουμε ιδέες για πολλά θέματα απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας και της υγείας. Θέλουμε να βοηθήσουμε όσους χαράσουν πολιτική και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να επωφεληθούμε όλοι. Η πρώτη κοινή διάσκεψη έγινε στο Λουξεμβούργο το 1998 και χαίρομαι που συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ετοιμάσουμε την 7η κοινή διάσκεψη σε ένα χρόνο από τώρα εδώ στις Βρυξέλλες. Εχθές συνάντησα τους κυρίους Κούς Ρισελ και τον κύριο Αμίντο Σίλβα για να κάνουμε κάποιες κοινέ εργασίες και μαζί θα προχωρήσουμε τις κοινέ μας εργασίες. Ελπίζουμε να έχουμε μια ακόμα επιτυχή κοινή διάσκεψη και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε στον τομέα αυτό. Μετά από την κοινή μα συνεδρίαση Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βοστόνη, ο οργανισμό μου εδεσμεύεται ακόμα περισσότερο στη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση OSHA και χαιρόμαστε που ε, ε, ενισχύουμε του δεσμού μα. Ένα τομεί ε, στον οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε είναι και η πρόληψη του εργασιακού καρκίνου. Παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε επαρκεί μελέτε, είμαστε βέβαιοι ότι σκοτώνονται χιλιάδε άνθρωποι καθημερινά από αυτό και ε, χαίρομαι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με τα θέματα αυτά. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον αμίαντο και να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε για να έχουμε και όρια έκθεσης ε, για άλλα γνωστά καρκινογόνα στοιχεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν να αντικαταστήσουμε καρκινογόνες ουσίες και να αναπτύξουμε και μηχανισμούς ελέγχου για αυτές τις οποίες δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα εργασιακού καρκίνου και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και είναι χρόνιες. Ε, συνάντησα ε, και τον Γκέρ Ντάνσετ από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Ουσιών ε, για να συζητήσουμε πώς μπορεί να βοηθήσει το ριτς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Εν τω μεταξύ, στι ΗΠΑ θα υιοθετεί ε, σύντομα ε, μία ενιαία παγκόσμια προσέγγιση για τους ε, κινδύνους εργασίας, για να μειώσουμε τους χημικούς κινδύνους, να μειώσουμε ε, τα προβλήματα για τους εργαζομένους και να διευκολύνουμε το εμπόριο. Πράγματι, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συμφωνούν ότι η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας και η αντιμετώπιση των χημικών παραγόντων είναι μεγάλη πρόκληση. Η θέση του οργανισμού μου είναι απλή. Πιστεύουμε ότι ε, η υπεύθυνη θέση οποιοδήποτε παραγωγού και εξαγωγέα επικίνδυνων υλικών θα πρέπει να ε, είναι να υπάρχει κατάλληλη επισήμαση για τα προϊόντα αυτά. Στον 20ο αιώνα ασχολούμαστε να βρούμε λύσεις για τους κινδύνους στην εργασία, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα πρότυπα που μπορούν να δώσουν διαδικασίες ώστε να ε, αναχαιτιστούν οι κίνδυνοι αυτοί. Ε, τα παραδοσιακά μέτρα ωστόσο τώρα δεν έχουν δώσει τον απαραίτητο θετικό αντίκτυπο, δεν ήταν επαρκή. Έτσι λοιπόν κοιτάζουμε πώς θα εμπλέξουμε τους ίδιους τους εργαζομένους και τους εργοδότες, στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα πρέπει να αλλάξει κατά τέτοιο τρόπο η νοοτροπία σε σχέση με το χώρο εργασίας, ώστε και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συλλογικά να αντιμετωπίσουν του κινδύνου υγεία και ασφάλεια. Στι ΗΠΑ κοιτάζουμε να προωθήσουμε προγράμματα πρόληψη για του τραυματισμού και τι ασθένειε, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και την διαχείρισή του. Στι περισσότερε τι μεγαλύτερε και διακρατικέ εταιρείε, καθώ και στι ε, εταιρείε των ΗΠΑ, έχουν εφαρμοστεί τέτοια προγράμματα τα οποία έχουν επιτρέψει με την πρόληψη, με την πρόληψη να αντιμετωπιστούν οι τραυματισμοί, να σωθούν ζωέ και να μειωθούν τα κόστη. Το ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ μοιράζονται ένα κοινό όραμα. Τα προγράμματα πρόληψη πρόληψη είναι καθοριστικά για τη βελτίωση τη ασφάλεια και τη υγεία των χώρων εργασία. Πρόσφατα, με μια κοινή διάσκεψη ΗΠΑ με μια τριμερή ομάδα εργασία, ε, οι ευρωγνώμονε συζήτησαν το κατά πόσο μπορεί να βρεθεί συμφωνία για τα απαραίτητα αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ να αφήσουμε ένα, από, ένα θα πρέπει η μέχρι τώρα επιτυχή συνεργασία μα να είναι ένα παράδειγμα για το πώ τα εργαλεία αυτά εξυπηρετούν εργαζομένου και εργοδότε ώστε να εφαρμοστούν επιτυχώ τέτοια προγράμματα. Οι προσεγγίσει μα έχουν πολλά α, ε, κοινά. Τα στατηγικά δικά μας σχέδια μπορούν να επιτρέψουν επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να ε, διαμορφώσουμε κοινέ προτεραιότητε και πρωτοβουλίε. Δεν είναι εκπληκτικό ότι κάθε φορά που συναντιούνται οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρουμε να ανταλλάξουμε ιδέε, να μοιραστούμε απόψει για τα προβλήματά μα, να βρούμε λύσει. Οι προοπτικέ μα και οι συνθήκε των εργαζομένων μα μοιάζουν, καθώ μοιάζουν ε, οι οικονομίε και οι κοινωνίε μα. Επίση, υπάρχει και η πολυεθνική διάσταση για τι οικονομίε και του εργαζομένου μα. 10% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα απασχολούνται από ε, εταιρείε Αμερικανική ιδιοκτησία και το αντίστροφο ε, σε ένα ποσοστό 10%. Υπάρχει πλέον παγκοσμιοποίηση στο εμπόριο και την απασχόληση. Και ε, η προστασία των εργαζομένων αυτή δεν έχει παγκοσμιοποιηθεί σε, παρόμοιο βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι ΗΠΑ να δούμε πώ μπορούμε να έχουμε περισσότερη προστασία για του εργαζόμενου σε παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στο σπίτι του, στι οικογένειέ του ασφαλεί μετά την εργασία του. Και θα πρέπει τα θέματα θέματα αυτά να αποκτήσουν εργασιακό χαρακτήρα. Η ασφάλεια και η υγεία θα πρέπει να απασχολούν και στι συζητήσει περί οικονομικών του ηθήνοντε. Δεν πρέπει λοιπόν εδώ να ξεχάσουμε και ένα άλλο σοβαρό ερώτημα. Πώ μπορούμε να παράγουμε περισσότερα καταναλωτικά αγαθά για την Ευρώπη και τι ΗΠΑ, εξασφαλίζοντα τι ευθύνε των εργαζομένων και την προστασία του στι αναδυόμενε επίση βιομηχανικέ ε, ε, δυνάμει θα πρέπει οι καταναλωτές, ε, τα προϊόντα των εργαζομένων να μπορούν να τα λαμβάνουν χωρίς να έχουν τεθεί σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια. Έτσι λοιπόν στη Διατλαντική Εβδομάδα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την διατλαντική σχέση μεταξύ των κρατών μας και για την κοινή δράση μεταξύ, Αμερικανικής, ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, στην ε, περίοδο της οικονομικής ε, κρίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εμπορικές ροές, την απώλεια θέσεων εργασίας, το πόσο έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση επιχειρήσεις και εταιρείε και το πόσο λιγότερο προστατεύονται αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν σε, μια σε ένα παγκοσμιοποιημένο χώρο εργασίας δεν μπορούμε να έχουμε περιτέ ή αναποτελεσματικέ βιομηχανικέ λύσει και τίποτα δεν είναι χειρότερο από του εργαζόμενου που ασθενούν, τραυματίζονται ή ε, πεθαίνουν λόγω προβλεπόμενων κινδύνων. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε την απαραίτητη ρυθμιστική προστασία για του εργαζόμενου και να ε, αποφύγουμε του περιττού τραυματισμού ή τι ασθένειε. Θα πρέπει τα μέτρα μα να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικά και οι εργαζόμενοι πιο παραγωγικοί, ε, πιο καινοτόμα τα μέτρα που χρησιμοποιούμε και όλο το περιβάλλον πιο ανταγωνιστικό και πιο επικερδέ. Οι αποδείξει που έχουμε από την πείρα μα είναι σαφή. Οι ρυθμίσει δεν καταστρέφουν τι θέσει εργασία, αλλά εμποδίζουν τι ε, θέσει εργασία ώστε να σκοτώνουν του ίδιου του εργαζόμενου. Σε αυτού του καιρού ανταγωνιστικότητα και προκλήσεων, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή χρειάζονται ο ένα τον άλλον περισσότερο από ποτέ. Μπορούμε λοιπόν και από τι δύο ε, πλευρέ του Ατλαντικού να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, πιστεύω, και να βελτιώσουμε το περιβάλλον σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι, ε, αυτή είναι κατάλληλη στιγμή για αισιοδοξία, για να είμαστε φάνταστη, να δείξουμε τόλμη και το πόσο μπορούμε να αναλάβουμε δράση. Ε, αρετές που χαρακτηρίζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ λοιπόν ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δέσμευσή του για την εργασιακή ασφάλεια και υγεία. Και επίσης είναι σοβαρή εδώ η συμβολή και του δόκτωρα Τάκαλα, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά, ε, του Διευθυντή μάλλον για τα θέματα αυτά, στο Διεθνές Πάνελ για τον ε, Επαγγελματικό Βίο. Εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα διεθνές δίκτυο ε, συνεργατών, ώστε να προωθήσουμε τις βελτιώσεις στο χώρο εργασίας και να μειώσουμε τις ασθένειες και τους τραυματισμούς χάρη και στη δική του συμβολή. Ελπίζω λοιπόν ότι η νέα διευθύντρια του Οργανισμού για την ε, Εργασία και Ασφάλεια και Υγεία, κυρία Λάτσεκ, θα επιτρέψει να είναι ακόμη παραγωγικότερη η συνεργασία μα, η συνεργασία των δύο οργανισμών και στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν η Διατλαντική Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτειών να αναλάβει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση αυτών των διεθνών προβλημάτων. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Our first uh, question is uh, Mrs. Pani Przewodnicząca. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ κύριο Μιχαήλ, για τη θαυμάσια του παρουσίαση. Ε, είδατε ότι σας χειροκρότησαν τόσο πολύ. και στα δικαιώματα των εργαζομένων και αναφερθήκατε και στην ευθύνη. Αλλά η ευθύνη είπατε ότι είναι η ευθύνη των εργοδοτών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε ότι ένας εργαζόμενος είναι αρκετά υπεύθυνο, έχει ε, επίγνωση ότι η εργασία θα πρέπει να την εκτελεί με υπευθυνότητα για να μην αναλαμβάνει κινδύνους ούτε για τον αυτό του ούτε για την επιχείρηση και να μην διατρέχει καθένα κίνδυνο. Όσον αφορά την επίγνωση αυτή των εργαζομένων, όσο πάει και το επίπεδο της μειώνεται. Γιατί θεωρούν ότι έχουν μόνο ευθύνε, μόνο συγγνώμη δικαιώματα και καμία ευθύνη. Κάτι άλλο. Η Μεγάλη Βρετανία ε, δημοσίευσε πληροφορίες για την αμνησία λέγοντας ότι οι νέοι 20-40 ετών υποφέρουν από την κατάσταση αυτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης μελέτες έρευνες κατά πόσον το άγχος έχει επιπτώσεις στην αμνησία. Thank you. Uh, Mr. follow... Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας και μετά η κυρία Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. The David Michael. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο David Michael για αυτό που μας είπε μόλις τώρα. Εδώ και πολύ καιρό ακούμε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού μόνο φωνές ε, και κριτικές, αλλά τώρα ακούμε ότι θέλει να είναι εταίροι μας για ένα καλύτερο κόσμο. Και αυτή η έκκληση με κάνει ευτυχισμένο γιατί πιστεύω ότι έχουμε πολλές ικανότητες, έχουμε πολλές ευθύνες και η μεν και η δε. Θα πρέπει από κοινού να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουμε στον οικονομικό τομέα και είναι καλό να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε ο κόσμος στον οποίο ζούμε να γίνει καλύτερος. Σας ευχαριστώ λοιπόν γιατί μας είδε πραγματικά μία πνοή νέου ανέμου, μία ελπίδα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Είμαστε πάλι πολύ ικανοποιημένοι γιατί θεωρούμε ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου, στην αρχή βρισκόμαστε και όσο πάει ενδυναμώνονται οι προσπάθειες στην έκτη διάσκεψη το επόμενο έτος θα μπορέσει νομίζω να αναπτυχθεί αυτό το θέμα. Περιμένουμε πολλά από τους Αμερικανούς φίλους μας και νομίζω ότι πραγματικά οι παραδοσιακοί μέθοδοι δεν αρκούν γιατί όσο πάει προχωράει η παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν να αντιμετωπίσουμε τις ε, παγκοσμιοποιημένες ασθένειες, αν θέλετε, των επιχειρήσεων. Τελειώντας, θα ήθελα να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία και να ε, ελπίσω ότι δεν είναι η τελευταία φορά που ερχόσαστε να μας επισκεφτείτε και όταν ξανάρθετε στις Βρυξέλλες ελπίζω να κάνει και καλύτερο καιρό. Παρόλο που δεν είναι ποτέ πολύ καλός και ο καιρός στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ για αυτή σας την ε, παρέμβαση, διότι θυμόμαστε έτσι ότι το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί πλέον θεμελιώδης δικαίωμα. Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τις συνθήκες εργασίας τους ε, διασφαλισμένες, εγγυημένες, η υγεία τους, η ασφάλειά τους να... και η αξιοπρέπεια τους πάνω απ' όλα να είναι ε, εγγυημένα στοιχεία. οι δυσκολίες που έχει κανείς στην εργασία, ε, το άγχος, η παρενόχληση και ούτω καθεξής είναι φαινόμενα που μας κάνουν να σκεφτόμαστε κατά πόσο είναι σωστά διοργανωμένη η εργασία, οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Μιλήσατε για, τον, για την χρηματοοικονομική, την ε, δημοσιονομική κρίση. Όλα αυτά αναστατώνουν την αγορά και εξαπλώνονται όλο και περισσότερο οι επισφαλεί μορφές απασχόλησης. Είναι η κλασική αντίδραση του να λέμε ότι υπάρχουν πολλές μα πολλές ε, μικρές συμβάσεις και οι επιχειρήσεις είναι δικαιολογημένες που δεν αναλαμβάνουν δράση για να συλλογικά να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα όπως το κόστος των ατυχημάτων και των ασθενειών που φτάνουν το 5,9 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε κόστος. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα, μια νέα νοοτροπία στις επιχειρήσεις. Πρέπει να υιοθετήσουν ε, την ε, ευημερία των εργαζομένων του ως ανάγκη και να αναλάβουν τι απαραίτητε δεσμεύσει. Πρέπει λοιπόν εδώ να κρόσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση των ποσοστών καρκίνου. Καρκίνο που σχετίζεται με την άσκηση επαγγελματικών ε, καθηκόντων. Εδώ ο συναγερμός αυτός πρέπει να ηχήσει και για όλες τις χημικές ουσίες που αύριο θα βρεθούν στην αγορά. Να θεσπίσουμε λοιπόν μια πραγματική αρχή πρόληψης και προφυλαξής, να εφοδιαστούμε με τα μέσα, ώστε όλες αυτές οι ουσίες να υπόκεινται σε μια διαδικασία αδειοδότησης. Ε, έχετε δημοσιεύσει ένα βιβλίο. Εγώ ως εισηγήτρια έχω παρακολουθήσει την σχετική επικαιρότητα με μεγάλη προσοχή καθώς και τις εργασίες σας. Ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαιτέρως που προσήλθατε στην Επιτροπή μας. Uh, Ευχαριστώ. Προς τόσο, σου για να απαντήσετε να υποβάλω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά τη σχέση ε, για την οδηγία... Ε, για την οδηγία που προσεχώς θα έρθει στην ε, Επιτροπή μας και να ξέρω πώς την αναμετήσετε στις είπα, υπάρχει ένας εθελοντικός ε, κώδικα συμποράφορας αυτή τη στιγμή. Θα ήταν όμως ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθεί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες όπως η οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και εκεί κάτι θα υπάρξει προσεχώς. Μήπως θα μπορούσαμε να μας δώσετε κάποια ιδέα το τι γίνεται στις ΗΠΑ ε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Και επίσης όταν συζητάμε το θέμα της συνεργασίας ε, και της πρόθεσης ε, παγκοσμίων πρωτοβουλειών, αργότερα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σε όλα τα θέματα, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς τοποθετήσετε εσείς σε πολλά αυτά τα θέματα. Έχετε το λόγο να απαντήσετε στι ερωτήσει. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί τόσο θερμή υποδοχή που μου κάνατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσει με τη σειρά που υποβλήθησαν. Το πρώτο, όσον αφορά τη σχέση των δικαιωμάτων και ευθυνών των εργαζομένων και των ε, στον τόπο ε, ε, ε, στην Αμερική ο νόμος λέει ότι θα πρέπει ο, ο εργοδότης να δώσει ε, όλες τις δυνατότητες ότι το περιβάλλον εργασίας να είναι ασφαλές. Δεν αναφέρονται τα δικαιώματα, δεν αναφέρονται οι υποχρεώσεις των εργαζομένων γιατί υποτίθεται ότι έχουν όλες τις δυνατότητες στα χέρια τους. Εμείς απαιτούμε ο εργοδότης να προσφέρει μια ασφαλή εργασία. Αν δούμε ότι τι κάνουν οι εργαζόμενοι και όχι τους όρους εργασίας, πολλές φορές χάνουμε τους λόγους ε, ατυχημάτων. Ένας εργαζόμενος πολύ εύκολο μπορεί να κάνει ένα λάθος. Και μπορούμε να πούμε επειδή έκανε ένα λάθος φταίει εκείνος για το ατύχημα. Ε, όμως δεν μπορεί να αποφύγει κανένας ε, ε, ένα λάθος στην καθημερινή του εργασία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να φροντίσει ούτως ώστε ένας λάθος να μην οδηγεί σε τραυματισμό. Εγώ για την αμνησία δεν ξέρω καμία έρευνα. Ενδιαφέρον το θέμα. Όταν γυρίσω στην ΣΥΠΑ θα το εξτάσω. Τώρα το θέμα της σχέσης παιδείας και εκπαίδευσης, βέβαια αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίζεται, να είναι μια δυναμική διαδικασία. Γιατί για να εργαστεί κανένα με ασφάλεια πρέπει να γνωρίζει του κινδύνου που απορρέουν από το υλικό με το οποίο εργάζεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέρκα για τα σχόλιά του και χάρηκα που είμαι τόσο Καλό δεκτό. Ε, Ξενόμητος του Υπουργού Εργασίας της ε, κυβέρνησης Ομπάμα, χαιρόμαστε πάρα πολύ να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Και σε εσά, ε, κυρία Τελή, τα σχόλια σα ήταν πολύ θετικά. Αναφερθήκατε στο θέμα της αξιοπρέφησης και της οργάνωσης της εργασίας. Οπωσδήποτε, η εργασιακή ασφάλεια και η υγεία εξαρτάται πάρα πολύ με την οργάνωση εργασίας, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί εκ των άνω. Πρέπει να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι. Πάντως χάρη, όταν ε, γίνεται ένα δυστύχημα, ε, ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους και τους εργοδότες να εξετάζουν τι, γιατί, πώς. Για να αποφευθούν λοιπόν οι τραυματισμοί, υπάρχει ένας πραγματικός Ειδικά ασφαλείς χώρους εργασίας θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Και αυτό βέβαια θέτει το θέμα ότι θα πρέπει να συνεργάζονται με κάθε σεβασμό οι μεν με τους δε. Και αναφερθήκατε επίσης στο θέμα των καρκίνων. Και είναι πολύ θετικό που συγκεντρώνεται στην Ευρώπη την προσοχή στο θέμα αυτό. Ο κ. Στάκαλα νομίζω θα αναφερθεί. Ε, το πρόγραμμα REACH δίνει πάρα πολλές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερωθούμε και εμείς και εργαζόμενοι. Περί τίνος προεκτός να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, ούτως ώστε ε, οι πληροφορίες ε, που προέρχονται από το σύστημα REACH να μπορούν να φτάσουν μέχρι τους εργαζόμενους που θα χρησιμοποιήσουν τις ουσίες αυτές. Κάτι άλλο. Η έκθεση των εργαζομένων ε, γίνεται συχνά μέσα στα πλαίσια του REACH και της ανάλογης νομοθεσίας της ΕΠΑ. Γιατί η έκθεση των εργαζομένων είναι το χειρότερο. Εγώ έχω εδώ μία καρφίτσα είναι ένα καναρίνι σε ένα κλουβί. Και ο λόγος αυτός είναι ότι οι εργαζόμενοι σήμερα είναι σαν τα καναρίνια που πέρανε παλιά στα ορυχεία οι, ε, εργάτες και όταν ε, δεν ήταν καλός ο αέρας στα ορυχεία ψόφαγε το καναρίνι και ο εργάτης ήξερε ότι υπάρχει κίνδυνος και ανέβαινε στην επιφάνεια. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι εργαζόμενοι έχουν τη χειρότερη έκθεση στις επικοινωνίες αυτές. Γίνονται πολλές μελέτες, ε, μελέτες για ζωά, αλλά παραδείγματο χάρη έχουμε το PPA που ε, η, τα πειράματα ανθρώπους αν θέλετε, οι έρευνες ανθρώπους γίνονται στους, εργα... στους εργαζόμενους στην Κίνα έχουμε κάποια τέτοια μελέτη που δείχνει τα αποτελέσματα ότι χάνεται τη δυνατότητα να παρουργήσει οι εργαζόμενοι αυτοί. Λοιπόν, με τα αποτελέσματα του θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και σε εσά και στις είπα Τέλος κυρία Πρόεδρε. Οι ε, ε, ε, τα μειοσχελετικά προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Τι στάνταρ διαδικασίε είναι όμω πολύ αργέ και δύσκολε. Έτσι δεν έχουμε εμεί σωστά πρότυπα για το θέμα αυτό, το να προστατεύουμε του εργαζόμενου από αυτέ τι παθήσεις. Ξέρω ότι κινείστε προ την κατεύθυνση αυτή και είμαι πολύ αισιόδοξο και υποστηρίζω πραγματικά τι προσπάθειές σα. Για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν ξέρω. Ε, μπορώ να σα δώσω όμω πληροφορίε, αν θέλετε, αλλά δεν έχω τα στοιχεία στα χέρια μου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ εξ ονόματος της Επιτροπής μας να σας πω ότι πρόκειται για μια πολύ καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ να μας απευθύνετε το λόγο σήμερα και αν θέλετε να παραμείνετε για το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη με τα χαράς. Κατανοώ βέβαια ότι μπορεί να έχετε και άλλες υποχρεώσεις και να πρέπει να φύγετε. Προχωράμε λοιπόν απευθείας στην έκθεση της ε, Καρή Μαντελή όπου θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας. Πριν ε, δώσω το λόγο στην Καρή Μαντελή, θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Έξι ως 8 λεπτά ο καθένας σας. Αντώνιο Καμαρότο, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης καταρχάς και μετά οι υπόλοιποι στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και 6-8 λεπτά. Έχουμε μία παρουσίαση με διαφάνειες. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ σήμερα. Χαίρομαι που μπορώ να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορώ να σας παρουσιάσω το ζήτημα αυτό, το οποίο αφορά την προετοιμασία της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης ε, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια και την Υγεία στον χώρο της εργασίας. Η αρχική μου παρουσίαση σήμερα αφορά την εφαρμογή της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και κάποιες πτυχές των βασικών εξελίξεων στο θέμα αυτό ιδίως ε, κάποιες προτεραιότητες τις οποίες εξετάζουμε για το για την επόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της ε, απασχόλησης. Ακούσαμε μόλις ε, τώρα ότι γνωρίζουμε όλοι το μέγεθος και τις επιπτώσεις των εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών και από πλευράς ε, προβλημάτων για τους ανθρώπους αλλά και τις οικονομικές συνέπειες παγκοσμίω. Μόλις ακούσαμε τον συνάδελφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο οποίος έχει τις ίδιες ανησυχίες με μας ε, για το θέμα αυτό. Η ανάπτυξη της κατάλληλης απάντησης επί του θέματος λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και να ανταλλάζουμε και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι σημαντικοί παράγοντες στον τομέα ε, εθνικά και ευρωπαϊκά ιδρύματα, ενδιαφερομένους ε, και εμπειρογνώμονες σε όλα τα ε, επίπεδα. Μας χαροποιεί λοιπόν ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, συνθήκες εργασίες ε, και την αντιμετώπιση ατυχημάτων και ασθενειών στα κράτη-μέλη και σήμερα ε, το θέμα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι σίγουρα μία από τις πιο ανεπτυγμένες πτυχές της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και ένας από τους βασικούς πυλώνες του λεγόμενου ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τις προκλήσεις ε, με τις οποίες ε, είμαστε αντιμέτωποι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ε, και για τους ανθρώπους και για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, προσπαθεί να διαφύγει της κρίσης και να ξεκινήσει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά αντιμετωπίζει ακόμα βεβαιότητες ε, για το κατά πόσον θα τα καταφέρουμε. Επειδή ακριβώς λοιπόν είναι τόσο δύσκολο το υπόβαθρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσίασε το 2010 μια νέα στρατηγική ατζάντα, τη λεγόμενη ε, Ατζέντα Ευρώπη 2020, που στόχο έχει να κάνει μια διαθερωτική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ο στόχος, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι να διαμορφώσουμε το μέλλον ε, των χωρών μας ώστε σε 20 χρόνια να έχουμε περισσότερη καινοτομία, λιγότερες περιβαλλοντικές ζημίες και ένα κατάλληλα εξοπλισμένο από πλευράς δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό. Για να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε κατάλληλο ρόλο θα πρέπει να έχουμε και κατάλληλες πολιτικές. Για να μειώσουμε τον αριθμό των ατυχημάτων και των ασθενειών στο χώρο της εργασίας, ε, που είναι στόχος ε, αφεαυτός, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις για το μέλλον. Τα ακούσαμε άλλωστε και από αρκετούς από τους προλαλήσαντες. Θεωρούμε όμως και εμείς ότι η βελτίωση των πολιτικών ε, για την ασφάλεια στην υγεία και την υγεία στον χώρο της εργασίας ε, σημαίνει ότι θα βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, θα έχουμε λιγότερες απουσίες και θα έχουμε και περισσότερες ε, και καλύτερες δυνατότητες ευημερίας είναι σαφές ότι για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσαρμόσουμε και τις πολιτικές μας τις αλλαγές οι οποίες ε, συμβαίνουν στο χώρο της εργασίας. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια όπως βλέπετε έχω ένα κατάλογο αυτών που θεωρούμε τις πιο σημαντικές πτυχές ε, των αλλαγών. Καταρχάς τις δημογραφικές αλλαγές, ε, διότι πλέον αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 50 ετών και αναμένεται ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο ενεργός πληθυσμός στην Ευρώπη. Επίσης, η μετατροπή των μορφών εργασίας, ε, που είναι πολύ σημαντικό διότι ε, η οικονομία μας θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανταγωνιστικές πιέσεις παγκοσμίω και θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες οργανωτικές δομές, ε, όλο και περισσότερο μεταβατικούς εργαζόμενους μεταξύ διαφόρων θέσεων εργασίας και ε, άτυπες μορφές εργασίες, ε, όπως για παράδειγμα η μερική απασχόληση που βλέπουμε ότι ολοένα αυξάνονται. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνέπειες των τεχνολογικών καινοτομιών που σημαίνει ότι έχουμε νέες διαδικασίες και νέα προϊόντα και φυσικά και νέους παράγοντες κινδύνου. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε και αυτή άλλωστε είναι και η πρόθεση και το πνεύμα της στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020 ότι χρειαζόμαστε καλύτερη ποιότητα ε, θέσεων εργασίας και συνθήκες εργασίες και είναι βασικός παράγοντας για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαρτώνται από την ε, επέκταση του εργατικού δυναμικού για την επιβίωσή τους και φυσικά θα πρέπει να έχουμε ένα ε, περιβάλλον εργασίας με ασφαλέστερες ε, συνθήκες εργασίας και αυτό είναι ζωτική σημασία. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε την ποιότητα εργασίας ε, για να μπορέσουμε να έχουμε ε, καλύτερη ε, εργασία. Έχουμε πιο εντατικές, πιο απαιτητικέ ε, θέσει εργασία πλέον. Ε, οι περισσότεροι εργαζόμενοι περνούν πολύ πιο εύκολα από τη μια δουλειά στην άλλη από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές ε, ε ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε πολιτικές για να έχουμε μια βιώσιμη εργασιακή ζωή και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες κάποιου σε όλο τον εργασιακό του βίο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την ποιότητα εργασία, διότι αυτό είναι φυσικό συμπλήρωμα τη δημιουργία θέσεων εργασία και καταλήλων προποθέσεων για μόνιμε θέσει εργασία και παραγωγικότητα. Βεβαίω, για να έχουμε την πλήρη εικόνα της σημερινή κατάστασης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιου πιο παραδοσιακού δείκτες που δείχνουν πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις στην κατάσταση στο συγκεκριμένο τομέα και τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Για παράδειγμα το γεγονός ότι έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα ε, ε ετησίως άνω των 5.500 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ε, στοιχεία που έχουμε από μια πρόσφατη δημοσίευση της Eurostat και βλέπετε επίσης ότι το 2007 που είναι το έτος αναφορά για τα στατιστικά στοιχεία αυτά Είχαμε πάνω από 5.500 ε, θανάσιμα ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο χώρο της εργασίας. Ένα περίπου 3% των εργαζομένων είχαν ένα ατύχημα στο χώρο της εργασίας και επομένως κατά συνέπεια απουσία άνω των τριών ημερών. 8,6% των εργαζομένων ε, αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα υγείας που σχετιζόταν με την ε, ε, εργασία, που σημαίνει ότι έχουμε περίπου 23 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να σας πω άλλα στοιχεία, τα βλέπετε και εδώ στη διαφάνεια. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα για το λόγο αυτό, το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική της ε, για την παραγωγικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, όπου θέλουμε να προάγουμε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και να έχουμε και τη δυνατότητα να προάγουμε τον την ολοκλήρωση των, ε, της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο της εργασίας και σε άλλους τομείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε και μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της στρατηγικής αυτής, η οποία προέκυψε από μια μακρά διαδικασία διαβούλευσης που έγινε το 2010 και τα βασικά συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας είναι σαφή κατά την άποψή μας. Καταρχάς θεωρούμε ότι παρά τις πολύ σημαντικές αλλαγές οι οποίες ε, έγιναν στην Ευρώπη από το 2007, ιδίως οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η στρατηγική εξακολουθεί να είναι ε, η πλέον κατάλληλη και ο βασικός πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης ήταν να μειώσουμε τον ε, αριθμό των ατυχημάτων και επιτέθη ο στόχος ε, κατά σημαντικό βαθμό γιατί είχαμε μείωση κατά 25% των ατυχημάτων και των δυστυχημάτων στον χώρο της εργασίας. Φυσικά η τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής ε, θα μπορέσει να γίνει όταν θα έχουμε τα στοιχεία για το έτος αναφοράς 2012. Προς το παρόν όμως έχουμε ε, κάποια στοιχεία όσον αφορά τις τάσεις ε, τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της στρατηγικής που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση μείωσης ε, που συσχετίζεται και με ε, δεδομένα που εξετάσαμε για μια μακρότερη περίοδο των τάσεων των 10 ετών. Θα πρέπει βέβαια να κάνουμε πολλά ακόμα στη διάρκεια της τρέχουσας στρατηγικής. Έχω εδώ ένα κατάλογο για κάποιες από τις προτεραιότητες. Καταρχάς ε, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε την απλούστευση και την επικαιροτησποίηση της κείμενης νομοθεσίας ε, μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας 2004-40 για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και μία πρόταση για μία νέα οδηγία η οποία εγκρίθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων προσφάτως και πλέον είναι στη διαδικασία διαβίβασης ε, των νομοθετικών σωμάτων. Μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία που αναφέρθηκε νωρίτερα αφορά τη νέα οδηγία για τα εργονομικά στοιχεία Έχουμε και τα πρόσφατα αποτελέσματα της πρώτης διαδικασίας εφαρμογής ε, για την ε, στρατηγική για ε, των εργασιακών κινδύνων και της ασφάλειας και της υγείας. Θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε κοινά εργαλεία παρακολούθησης για την εφαρμογή των μελλοντικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα και βεβαίως ε, κατ' εξίσου σημαντικά θέλουμε να κάνουμε και τελικές αξιολογήσεις της τρέχουσας στρατηγικής και θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα περίγραμμα της μελλοντικής στρατηγικής για την περίοδο ε, μέχρι το 2020. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευρεία διαβούλευση εν εξελίξη η διαδικασία στόχο έχει επίσης να εντοπίσει και τις προτεραιότητες ε, για την στρατηγική παρακολούθηση, ε, η οποία θα πρέπει να συνάδει και με τη στρατηγική ε, για το 2020 και την περίοδο 2013-2020. Βεβαίως η νέα στρατηγική θα μας δώσει και το πολιτικό πλαίσιο για τη βελτίωση των της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο της εργασίας και θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει και τον οδικό χάρτη ώστε να έχουμε και την κατάλληλη εφαρμογή και την ε, ε, συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Αυτά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας παρόλο που ξεπεράσατε λίγο το χρόνο. Ο κύριο Στάκαλα τώρα. Εάν μπορούσατε να παραμένετε εσεί τουλάχιστον στα όρια του χρόνου, έξω με 8 λεπτά. Σα αφήνω να συστηθείτε μόνο σα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, μέλη του ε, Κοινοβουλίου, φίλοι και προσκεκλημένοι. Με αφορμή και την προηγούμενη συζήτηση που έγινα, μου πολύ αυτό που είπε ο Ντέβιντ Μάικλς ότι οι ρυθμίσεις δεν σκοτώνουν την απασχόληση, την εργασία, αλλά εμποδίζουν την εργασία, τις θέσεις εργασίας από το να θανατώνουν του εργαζομένου. Εγώ λοιπόν υπήρξα διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και συμφωνώ πολύ με αυτή τη δήλωση. Ε, κάθε χρόνο στην Ευρώπη 168.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους για εργασιακούς λόγους. Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός είναι κάπως αυξημένος. Όσο αυξάνονται τα ατυχήματα, τόσο τείνουν να, να μειώνονται οι ασθένειες. Επίσης, 20 είναι Πολλοί μάλλον ε, οι ασθενείς στην Ευρώπη που χάνουν το, τη ζωή τους λόγω διαφόρων μορφών καρκίνου και τον αναφέρω αυτό λόγω, ε, λόγω των εργασιών των σχετικών του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι πολλά τα ατυχήματα που επίση συμβαίνουν στην ε, διάρκεια της εργασίας. Επτά εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως, εργαζόμενοι ετησίως, και περίπου 20 εκατομμύρια εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι έχουν προβλήματα σχετικά με την υγεία τους. Αυτά μας τα λένε και οι ρυθμοί της Eurostat. Το είπε και ο συνάδελφός μου προηγουμένως. Είναι πολλοί οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να ασκήσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους. Πέραν λοιπόν του ανθρωπίνου κόστους, πρέπει να ασχοληθούμε και με το οικονομικό κόστος. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις γι' αυτό. Οι Αυστραλοί υπολογίζουν 5,9 του ΑΕΠ τους. 5,9%. Εμείς δεν έχουμε ακόμη ακριβή στοιχεία, αλλά θα τα επεξεργαστούμε στον οργανισμό μας και θα τα ετοιμάσουμε για το χρόνο. Επιπλέον, και αυτό είναι το σημαντικότερο, υπάρχουν απώλειες λόγω ε, αναπηριών των εργαζομένων που δεν μπορούν να φτάσουν την ε, ηλικία συνταξιοδότησης ή ε, υπάρχουν συστηματικές απουσίες. Αναγκάζονται να φύγουν νωρίς λόγω αδυναμιών ή αναπηριών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές δαπάνες σε εθνικό επίπεδο. Τα καλά νέα είναι ότι τα ατυχήματα μειώνονται στην Ευρώπη. Όμως άλλες πτυχές της ποιότητας της εργασίας όπως η πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση, την κατάρτιση δεν βελτιώνονται. Τι είναι λοιπόν το σημαντικότερο που θα πρέπει να σημειώσουμε. Εάν δούμε ότι έχουμε μηδενική αύξηση στον πληθυσμό και τις μειώσεις ε, στον αγορά εργασίας, στον πληθυσμό εργασίας, βλέπουμε να υπάρχει αύξηση στο συνταξιδοτικό όριο τα τελευταία 7 με 10 χρόνια. Η εργασία σε διάφορα είδη, σε διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων έχουν περισσότερες μειοσκελετικές ασθένειες. Επίσης ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και επιβαρύνσεις και υπάρχει και μεγαλύτερη έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και βιολογικού παράγοντες. Για παράδειγμα, στον τομέα τον υγειονομικών ή της κομματικής. Εδώ υπάρχει ένας σημαντικός ρόλος που μπορεί να διδεματίσει η τη κομμωτικη εδω υπαρχει ενας σημαντικος ρολος που μπορει να διαδραματίσει η ευρωπαικη ενωση για τους νεότερους, κάτω των 28 και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της γυρέσας του πληθυσμού. Συνήθω οι νέοι όμως αποσχολούνται σε επικίνδυνου κλάδου όπως τη γεωργία ή τι οικοδομές. Μπορεί να έχουν προβλήματα και στην κατανόηση της γλώσσα που χρησιμοποιείται προκειμένου να αναλάβουν πλήρω τις ευθύνε τους για την υγεία και την ασφάλειά τους. Αλλά και ο πληθυσμό ο γυράσκει. Όσοι πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκουν σε μια γενιά που όλο ένα και κλείπει. Οι εργαζόμενοι που θα συνταξιδοτηθούν σε 20 χρόνια θα έχουν συρρυκνωθεί ως ομάδα πληθυσμιακή έτη περαιτέρω μέχρι το 2040. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με ασθένειες εργασιακές οι οποίες είναι πηγή των προβλημάτων. Οι μειοσκελωτικές διαταραχές, υπόνοι στην πλάτη, πόνοι στο πάνω μέρος του σώματος, είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Η βιωσιμότητα λοιπόν στην εργασιακή ζωή είναι πολύ σημαντική. Είναι λίγοι χειρονάκτες που πιστεύουμε ότι θα φτάσουν στα 60 να κάνουν με την ίδιο τρόπο την εργασία τους. Σε σύγκριση λόγου χάρη με συναδέλφους τους στον σε, το, στον τομέα των υπαλληλικών. Επίση, είναι πολλοί εκείνοι που εργάζονται σε μερική απασχόληση, ιδίω οι γυναίκε ω αυτοπασχολούμενε, σε μικροεταιρείε ή με πολλέ ε, μικροδουλειέ ταυτόχρονα. Το θέμα είναι πώ θα εξασφαλίσουμε σε αυτού του εργαζόμενου την κατάλληλη εκπαίδευση. Πώ θα καλύπτονται από μέτρα πρόληψη. Πώ θα παρακολουθείται η υγεία του. Πώ θα συλλέγουμε δεδομένα για την κατάσταση τη υγεία και τη ασφαλεία του. βλέπουμε συνεχώς να εξαπλώνεται ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα όλων των ε, θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει και στενά να παρακολουθούμε τον κίνδυνο ατυχημάτων που γνωρίζουμε καλά και την έκθεση σε παραδοσιακούς όπως λέγονται τομείς. Να, είμαστε, να έχουμε επίγνωση για την υγεία και την ασφάλεια και τους ε, τις απειλές που αντιμετωπίζουν στον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πάντως, σημαντικά αίτια της απουσίας από την εργασία ε, πολλές φορές έχουν να κάνουν με μειοσκελετικές διαταραχές όπως τα προβλήματα πλάτης, αλλά και ψυχοκοινωνικά ε, ζητήματα όπως το άγχος, η κόποση, η κατάθλιψη που μπορεί να οδηγήσουν σε μακρόχρονες απουσίες για όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά περισσότερο μας ανησυχούν ε, για τις γυναίκες 135, νεαρές γυναίκες που πολλές φορές δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην εργασία τους. Αυτό πραγματικά είναι πολύ σχετικό σε ένα γυράσκοντα πληθυσμό που τίνει να ε, οδεύει περισσότερο προ την παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, ε, η ίδια, η, ο ίδιο ο εργασιακό πληθυσμό αλλάζει. Νέε απειλέ, νέε μορφέ έκθεση θα προκύψουν, διότι όλο και περισσότερο από το παραδοσιακό γραφείο ή το εργοστάσιο οι εργαζόμενοι θα τείνουν να μετακινούνται ε, στον χώρο των ασθενών ή να βρίσκονται στο σπίτι του ή να μετακινούνται διαρκώ. Δεν ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο θα είναι δυνατό για όλους να εργάζονται στο επίσημο συνταξιδοτικό όριο. Για 7 σήμερα έχουμε νωρίτερη, ε, πρώτερη συνταξιδότηση 7 με 10 χρόνια. Πιο νωρίς από ό,τι κανονικά προβλέπει το επίσημο όριο. Πάντως, ε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός και το Διεθνές Πάνελ στο οποίο σύντομα θα συμμετάσχω πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα του ε, βιώσιμου εργασιακού βίου. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η νομοθεσία, ε, η απαραίτητη καθοδήγηση, η τεχνική υποστήριξη θα δοθούν στους εργαζομένους που τις χρειάζονται. Ένα σημαντικό μέρος ε, της προσπάθειάς μας είναι να καταλάβουμε πώς η υγεία και η ασφάλεια είναι αντικείμενο μέρη καθημερινά στον εργασιακό χώρο. Ο προηγούμενος οργανισμός μου είχε αναλάβει ενεργό δράση εκπονώντας τη μελέτη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, επικεντρωνόμενο στην διαχείριση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και λαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στο να χρησιμοποιήσει ένα από τα πρώτα εργαλεία τα πολλά, που υπόσχονται πολλά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην υγεία και την ασφάλεια. Περισσότερες από 36.000 ε, συνομιλίες μας έδειξαν με τη μελέτη αυτή ότι ε, υπάρχει υψηλό επίπεδο ανησυχία μεταξύ των ε, Ευρωπαίων Εθνών για τα θέματα του εργασιακού άγχους, λόγου χάρη. Πρέπει να θυμόμαστε εδώ ότι το στρες, το άγχος μπορεί να προλαμβάνεται. Υπάρχουν σημαντικές εδώ αποκρίσεις και εδώ επιλεκτικά έχω σταθεί σε κάποια σημεία της μελέτης μας, τα οποία νομίζουμε θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε μελλοντικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλίες ε, με ένα εργαλείο ε, διαδικτυακής αξιολόγησης του κινδύνου, όιρα όπως ονομάστηκε, κάτι που θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλα κατημέλη, ήδη γίνεται αυτό σε έναν βαθμό, και να ε, υλοποιηθεί με τη βοήθεια των κοινωνικών εταιρών σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πρακτικό μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή πολλών εργαζομένων και να απλουστεύσουμε τις καθοδικατικές μεθόδους θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική που να μας επιτρέψει να ε, εξετάσουμε το θέμα αυτό σφαιρικά με προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων. Σας παρακαλώ λοιπόν, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα που υπάρχουν, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που προέρχονται από το παρατηρητήριο κινδύνων εργασιακών. Εδώ Βλέπετε, 20 με 30 χρόνια γίνεται ήδη μια προσπάθεια. Χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτέ τι πολύτιμε πληροφορίε όταν χαράζετε πολιτικέ για τι μελλοντικέ μα γενιέ. Και να θυμάστε ότι δεν αρκεί να εντοπίζουμε μόνο τα προβλήματα, ε, πράγμα που ήδη κάνουμε, αλλά πρέπει να προτείνουμε και λύσει. Πρέπει να είναι οι λύσει που προτείνουμε φιλικέ προ το χρήστη και να φροντίσουμε οι χώροι εργασία τη Ευρώπη να είναι πιο παραγωγικοί ο υγιεινό χώρο εργασία είναι καλό και για του εργαζόμενου και για τι επιχειρήσει. Και μια προσωπική παρατήρηση. Αυτή είναι η τελευταία μου συμμετοχή στι εργασίες τη Επιτροπή σα Θα συνταξιδοτηθώ το Σεπτέμβριο. Ήθελα λοιπόν να σα εκφράσω τη βαθιά μου γνωμοσύνη για την ε, καλοσύνη σα και για τη στήριξή σα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μεγάλη μου χαρά που συνάντησα σήμερα εδώ τον David Michaels. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί. Επίσης είμαι βεβαίως ότι η διεθνή συνεργασία θα παραμείνει εντατική, εύρωστη και Χαίρομαι που βλέπω ότι η Κρίστα Σέντλατσε, παρόλο που φοράει μικρότερο νούμερο παπούτσια από μένα, έχει αναλάβει αυτή την υπεύθυνη θέση. Και θα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από νέε προκλήσει. Χαιρετώ λοιπόν του καλεί μου φίλου και σα εύχομαι καλή τύχη για το μέλλον. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε και σε εσά, αγαπητοί και αγαπητέ βουλευτέ, συνεχίστε να μα στηρίζετε στι προσπαθίε μα. είμαι σίγουρη ότι θα σας άρεσαν τα χειροκροτήματα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε ξανά. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μίλτερ από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ καταρχήν που καλέσατε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας όταν εξετάζετε το θέμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και την έκθεση που θα προετοιμάσετε από αυτού. Θα σας παρουσιάσω το πώς συμβάλλει η Eurofound, ένας τριμερής οργανισμός από τις διεθνείς αρχές ε, και τους ε, ε, κοινωνικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμβολή, λέω, που προσέφερε ο οργανισμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Καταρχήν, η έρευνα για τους σώρους εργασία. που κάνουμε από το 90 ήδη και ε, αφορά ένα ε, αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 34 χώρες μάλιστα πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία σειρά ερωτήσεων για την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, τους όρους εργασίας γενικά. Η έρευνά μας αυτή επιτρέπει να δείτε τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα με την πάροδο του χρόνου. Να δείτε κατά πόσο υπάρχει πρόοδος ή επιστοχώρηση. Σας επιτρέπει να ε, αναγνωρίσετε τους παράγοντες κινδύνου και εξ αυτού Μπορούν έτσι οι διάφοροι παράγοντες να παρέμβουν. Είτε οι κοινωνικοί εταίροι ή η οι πολιτικοί. Και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε τρία-τέσσερα σημεία της έρευνάς μας συγκεκριμένα. Πρώτο σημείο. Η εντατικότητα της εργασίας. Η ένταση της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό όταν το λέμε αυτό, αναφερόμαστε στο ρυθμό της εργασίας. Το ρυθμό με τον οποίο είναι αναγκασμένοι να εργάζονται οι εργαζόμενοι. Ο ρυθμός αυτός της εργασίας αυξήθηκε τα 20 τελευταία χρόνια. Φαίνεται όμως ότι σταθεροποιείται σε υψηλό επίπεδο. Ο ρυθμός αυτός της εργασίας είναι ένας δείχτης και θα δούμε αργότερα ποιος είναι ο κίνδυνος. Μετά, οι φυσικές απαιτήσει στο χώρο εργασίας. Φυσικά, επίσης, σημαίνει να σηκώνει κανένα μεγάλα βάρη, να εργάζεται σε δύσκολες ε, θέσεις του σώματος, η χρήση της χρώση του χεριού αν θέλετε γενικά επαναλαμβανόμενα ακόμα και ο κόσμος της εργασίας σήμερα έχει αλλάξει δηλαδή λιγότερο στη βιομηχανία και στην γεωργία και περισσότερο στις υπηρεσίες. υπηρεσίε όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκε. Τρίτον, αυτονομία στον τόπο εργασία. Αυτονομία στον τόπο εργασία σημαίνει να μπορεί κανένα να παρέμβει στη μέθοδο εργασία, στη σειρά εργασίας ή στην ταχύτητα με την οποία εργάζεται. Η αυτονομία αυτή στον τόπο εργασία είναι ένα τρόπο για να μπορέσει να απτυχθεί μια ευημερία στον τόπο εργασίας. Να μπορούν έτσι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να έχουν τη δυνατότητα να αυτοδιοικούνται αν θέλετε. Η αυτονομία αυτή στον τόπο εργασίας παρέμεινε λίγο πολύ σταθερή. Δεν αυξήθηκε δηλαδή. Γενικά λέω, αλλά υπάρχουν και ομάδες κινδύνου. Δηλαδή ε, εκείνοι που εργάζονται χειρονακτικά που έχουν τη λιγότερη αυτονομία. Εάν η αυτονομία στον τόπο εργασία είναι ε, η προϋπόθεση της πρόληψης και μια που βλέπουμε ότι η ένταση και οι σωματικές απαιτήσει στον τόπο εργασία αυξάνονται Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση, αλλά ο έλεγχος της εργασίας παραμένει ο ίδιος. Και ο εργαζόμενος έχει λιγότερη αυτονομία. Αυτές οι πηγές δηλαδή άγχους αυξάνονται. Οι πηγές του να μην ελέγχει κανένας αυτό που κάνει. Οι σωματικές απαιτήσεις στον τόπο εργασία είναι η πηγή για, τους, για τα μειοσκελετικά προβλήματα. Και επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να παρουσιάσω και ένα άλλο σημείο όσον αφορά τον τύπο συμβάσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα. Οι συμβάσεις απεριορίστου χρόνου παραμένουν ο κανόνας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε με την ερευνά μας ότι οι συμβάσεις προσωρινής εργασίας αυξάνονται. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια τριγωνική κατάσταση. Ο εργαζόμενος, η επιχείρηση που τον χρησιμοποιεί και η μεσάζουσα υπηρεσία, η επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημειονεκτική θέση αυτός ο εργαζόμενος προσωρινά σε σχέση με εκείνο που εργάζεται πιο μόνιμα όσον αφορά και τα ε, ωφέλη του και όσον αφορά άδειες και τέτοια. Ο εργαζόμενος με περιορισμένο χρόνο εργασία είναι μια ομάδα κινδύνου γιατί δεν έχουν ασφάλεια για την θέση τους. Αλλά βλέπουμε επίσης από την έρευνά μας ότι υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία. Η νομοθεσία για την απογόρευση του καπνίσματος στον τόπο εργασίας οδήγησε τους εργαζόμενους να μην εκτίθενται τόσο πολύ στον καπνό όταν εργάζονται. Μακροπρόθεσμα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Η νομοθεσία λοιπόν μπορεί να συμβάλλει θετικά στην βελτίωση της κατάστασης. Η κοινοτική στρατηγική ανείχνευσε μια σειρά ομάδων κινδύνου, παραδείγματος χάνει μετανάστες. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενθαρρύνει τη μετανάσταση μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το εγγυάται η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία κυκλοφορίας. που υπάρχει ήδη στην συνθήκη της Ρώμης, στην ίδρυση δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά βάση, οι μετανάστες εργαζόμενοι δηλαδή ότι δεν είναι υπήκοοι στη χώρα που εργάζονται, καλύπτονται από την ίδια νομοθεσία και τις ίδιες συμβάσεις. Θεωρητικά. Στην πράξη τα πράγματα διαφέρουν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των υπηκών και των μη υπηκών, χωρίς να μπορεί κανείς να ανηγενικεύσει όμως. Παραδείγματος χάρη. Έρευνες για τους όρους εργασίας ε, εθνικών εργαζομένων στη Φιλανδία μας λένε ότι οι μη υπήκοοι έχουν συχνότερα ε, συμβάσει περιορισμένου χρόνου. Αν αναλύσει κανένας τα στοιχεία των δυστυχημάτων στο τόπο εργασία, ιδίω εξετάζοντας κάποιου τομεί επικίνδυνου όπως τι οικοδομέ, βλέπουμε ότι οι μη υπήκοοι εργαζόμενοι έχουν υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων από το εθνικό μέσο όρο. Η έρευνα για το εργατικό δυναμικό, η Labor Force Survey, μας λέει επίσης ότι κατά μέσο όρο οι υπήκοοι εργαζόμενοι παραμένουν περισσότερο χρόνο στον ίδιο εργοδότη από τους μη υπηκούς. Και αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί, πώς τους συμπεριφέρονται. Επίσης, είδαμε το θέμα της ε, απόκτησης υπηκότητας τα τελευταία χρόνια και τώρα έχουμε μια νέα κατηγορία και ο εργαζομένων που κινδυνεύουν. Δηλαδή έχουμε υπηκόους από που προέρχονται όμως από μια άλλη χώρα και που είναι θύματα καλυμμένης ε, διαφοράς ή διακριτικής μετα, Τώρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μελέτες μας κατέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι στις ΜΜΕ είναι λιγότερο καρά ενήμεροι όσον αφορά τους κινδύνους, ότι υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες και οικονομικές και γνώσεων της ΜΜΕ. Υπάρχουν βέβαια και πολύ ενδιαφέροντα θετικά παραδείγματα όπου οι ΜΜΕ συγκεντρώνουν τις δυνατότητές τους, ούτως ώστε από κοινού να μπορέσουν να ακτιμήσουν τους κινδύνους. Κατά γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, τόσο καλύτερα ενήμεροι είναι οι εργαζόμενοι οι μελέτες μας για τον κοινωνικό διάλογο και τις γνώσεις για την εργασία καταδεικνύουν ότι εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν την δυνατότητα να έχουν μέσα στην επιχείρηση κοινωνικό διάλογο βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από εκείνου που δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Κάτι που ενδιαφέρει όλους τους ε, ενδιαφερόμενους, εσείς όπως εσάς, είναι οι διάφορες μορφές συμβάσεων στον ίδιο τόπο εργασία. Όσο πάει και περισσότερο έχουμε την κατάσταση ότι στον ίδιο τόπο εργασία έχουμε 4-5 διαφορετικές μορφές εργασίας με διαφορετικές επιπτώσεις για τα άτομα αυτά. Και φυσικά και για την ατμόσφαιρα στον τόπο εργασίας. Το έχω αναπτύξει στο γραφτό μου έγγραφο και το έχετε στη διάθεσή σα. Τελευταίο σημείο κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει για τα θέματα αυτά να εργαστούμε περισσότερο τα επόμενα έτη. Ε, υπάρχει μία μελέτη που έκανε το Πνευσίου Λαβάλ στο Καναδά, στο Κεμπέκ και μας παρουσιάζεται εκεί ένα νέο φαινόμενο υψηλή και καλυμμένη πίεση. Όταν είναι στον τόπο εργασία οι άνθρωποι έχουν πιο υψηλή πίεση παρά όταν πάνε σπίτι τους ή μάλιστα αν πάνε στο γιατρό. Λοιπόν, αυτό το στρες, αυτό το άγχος μπορεί βέβαια να οδηγήσει να προέρχεται από την αβεβαιότητα της εργασίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και θέμα οργάνωσης εργασίας. Και συχνά της μη διαπραγμάτευσης για την αναδιοργάνωση της εργασίας. Οπωσδήποτε αυτό το θέμα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Α, τούτο λεχθέντον, κυρία Πρόεδρε, έχω να σας πω ότι το Ίδρυμα του Δουβλίνου είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσετε και με την, ε, το, την υπηρεσία του Βιλπάου και με την Κομισιόν και να εξεταστεί η στρατηγική για τη μείωση των ασθενειών και των δυστυχημάτων στον τρόπο εργασία που θα μπορούσε να προχωρήσει και μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς κάνοντας σχετικές έρευνες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Πριν ε, δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, η Κάρη Μαντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε για όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Να σας πω ότι κατά την άποψή μου ότι το να ε, συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία με 9 μόνο χιλιάδες χαρακτήρες είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα ζήτημα πραγματικά πολύ σημαντικό, μείζον προβληματισμός. Μία διαπίστωση τώρα, από το 2007 ως το 2012, που να δούμε πολύ κριτικό βλέμμα το όσο έχουν γίνει. Και θα πρέπει να είμαστε και πολύ φιλόδοξοι. Από την πλευρά των επικρίσεων λοιπόν, να πούμε ότι αν σήμερα διαπιστώνουμε μείωση του ποσοστού ατυχημάτων, ίσως αυτό έχει να κάνει και με την μείωση της απασχόλησης, των ποσοστών απασχόλησης και εργασίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τα πράγματα κατά πρόσωπο και να σκεφτούμε τι πρέπει να γίνει εδώ. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια προσέγγιση κατακαιρματισμένη. Η υγεία είναι ένα θέμα οριζόντιο. Και προσοχή πρέπει να δώσουμε στα ατυχήματα μεν, βεβαίω, αλλά το θυμήσατε κι εσείς, ο τελευταίος ομιλητής, ότι υπάρχουν και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Αυτοί οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι συνδέονται με το άγχος, τον σωματικό ε, πόνο, την ε, ε, παρενόχληση, την ανασφάλεια στο χώρο εργασίας και την κακή διοργάνωση της εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν. Μιλήσαμε προηγουμένω για μειοσκελετικέ ε, διαταραχέ, μιλήσαμε για βιολογικού και χημικού ε, κινδύνου. Αυτά έχουν όλα να κάνουν με το διοργάνωση τη εργασία. Τον, τη μέθοδο με την οποία διοργανώνεται δηλαδή. Και επίσης πρέπει να θυμόμαστε και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Εάν ε, επενδύσουμε σε αυτή τη διαδικασία, σίγουρα θα έχουμε μόνο ωφέλη να αποκομίσουμε. Διότι αν επενδύσουμε τώρα στην πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αυτό και την ευμερία μάλλον και την ευζοία των εργαζομένων θα επιτρέψει να καλλιεργήσουμε και θα μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις και κατά τρίτον λιγότερες δαπάνες θα σημαίνει και για την κοινωνία στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας. Πρέπει λοιπόν να γίνει προσπάθεια πραγματική Ιδίω σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων. Αυτό είναι ένα ζήτημα μείζων για την νέα αυτή στρατηγική. Πρώτα απ' όλα, οι κίνδυνοι είναι περίπλοκοι και πολύπλευρη. Επίση, υπάρχει περιπλοκότητα στον τρόπο λειτουργία των συστημάτων των κρατών μελών. Όμω, πρέπει να παραμένουμε φιλόδοξοι. Α πούμε, ο αμίαντο. Τι γίνεται με τον αμίαντο. Εδώ, ε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και διαδραμάτισαν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Στην έκθεσή μου τώρα, τι θα συναντήσει κανείς. Το έχω πει. Η έκθεση αυτή θέλω να είναι φιλόδοξη. Φιλόδοξη και χάρη στη δική σας τη συμβολή. Όμως θέλουμε να δώσουμε έμφαση και σε θέματα στα οποία για την ώρα δεν έχουμε ε, ε δεν είχε τύχει να έχουμε την ευκαιρία να αποδώσουμε αρκετή προσοχή. Πρώτα απ' όλα η εξωτερήκευση της ε, εργασίας είναι καθοριστική σημασία σε αυτό. Δηλαδή υπεργολαδία, εξωτερική ανάθεση. Αυτό πρέπει να το ε, επισημάνουμε με, με τη δέουσα προσοχή. Αφορά ε, επίσης και την εργασία ε, από απόσταση καθώς και την ευθύνη των εργοδοτών. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Ευθύνη των εργοδοτών στην συστηματική υλοποίηση πολιτικής πρόληψης. Όπως το είπατε και εσείς, Πρόεδρε, σας εύχομαι μάλιστα καλή συνταξιοδότηση. Αναφέρατε έναν αριθμό εκπληκτικό. 168.000 Ευρωπαίοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών. Εάν μιλήσουμε για αυτό το βακτηρίδιο το, στα αγκουράκια, δεκάδες θάνατοι και από αυτό αλλά για σκεφτείτε, μιλάμε για ατυχήματα στο χώρο εργασία. Ε, πρέπει να γίνει προτεραιότητα αυτό στην ευρωπαϊκή μα ε, ε, σειρά ε, προτεραιοτήτων. Στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πρώτο αίτιο λοιπόν θνησιμότητας στο χώρο εργασίας είναι και οι καρδιοαγκιακές παθήσεις και οι αναπνευστικές και τα ατυχήματα που όμως είναι ένα μικρό ποσοστό του συνόλου θανάτων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ολόκληρη πτυχή, ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην έκθεση για τα στατιστικά δεδομένα. Θα φροντίσω πραγματικά επισταμένος να ζητηθεί από την Επιτροπή να προβλέψει τα απαραίτητα στατιστικά εργαλεία ώστε να συλλέγονται στοιχεία ε, συστηματικώς για τα ατυχήματα αλλά και τις ασθένειες και το ποσοστό των εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε παράγοντες ε, βιολογικούς επικίνδυνες, χημικούς ή ψυχοκοινωνικούς κινδύνους ή που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και άρα επικίνδυνες. Έπειτα να σταθώ στο γεγονός ότι σήμερα χρειάζεται να είμαστε συνεπείς. Χρειάζεται συνοχή μεταξύ ευρωπαϊκού πλαισίου και εθνικών πλαισίων. Νομίζω ότι μόνο η ευρωπαϊκή δράση μπορεί να λειτουργήσει εφόσον είναι και εναρμονισμένη και πρέπει να είμαστε σαφείς. Άλλο πράγμα είναι η υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που για την ώρα θα πρέπει να απομένει να συνδυαστεί με τα εθνικά προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τι συμβαίνει σε επίπεδο κρατών μελών. Τι αξιολόγηση χρειάζεται εδώ και τι έλεγχος είναι αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Όλα αυτά σε πέντε σελίδες πολύ δύσκολα. Θα συμπεριληφθούν αλλά σας λέω χοντρικά τι θα βρείτε στη δική μου την έκθεση. Έπειτα η πρόληψη στο χώρο εργασίας, πρέπει να είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η εργασιακή ιατρική, η επιδημολογία, η τοξικολογία, η βιομηχανική υγιεινή, η ψυχολογία είναι τομείς που εμπλέκονται σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά μιλάμε για ένα πεδίο ευρύτατο. Επίσης, νομίζω θα το ξαναδούμε, η υλοποίηση της οδηγίας REACH είναι άκρα σημασίας είναι αναγκαία. Σήμερα χρειάζονται περισσότερε σχέσει συνεργασία μεταξύ τη πολιτική εργασιακή υγεία καθώ και των κοινοτικών πολιτικών αλλά και των εθνικών. Τέλο, να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντα ότι η κουλτούρα αυτή τη πρόληψη, η νοοτροπία υπέρ τη πρόληψη πρέπει να ενισχυθεί. Χρειάζεται ενδυνάμωση και πραγματικά να εκπροσωπούνται σωστά και οι εργαζόμενοι. Αυτό μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην υγεία τους, την ασφαλειά τους στο χώρο εργασία, ιδίω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν η εκπροσώπηση είναι και επίσημη, θέλουμε να υπάρχει σε κάθε περίπτωση γιατί είναι παράγοντας καθοριστικός για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασία. Πρωταρχικό είναι και ο ρόλο των ε, εποπτών εργασίας. Η εργασιακή ιατρική έχει να διαδραματίσει εδώ μια αποφασιστική συμβολή για την πρόληψη Και να θυμίσω εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουν στην κατάρτιση. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε ακόμη ε, σκληρά. Δεν είναι σημαντικό να ενημερώνονται μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και όλες οι επιχειρήσεις και οι μελλοντικοί ηθήνοντες, αυτοί που θα αναλάβουν στο μέλλον τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης και οι εργαζόμενοι σε ευάλωτη θέση και οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και οι μετανάστες και οι νέοι και οι γυναίκες οι γυναίκες μάλιστα που βρίσκονται σε ηλικία πρώτης μητρότητας, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι παρέχοντες υπηρεσίες, όλοι αυτοί είναι σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες. Επίσης, έχω διάφορα ζητήματα να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να διευρυνθεί η οδηγία που αφορά τους καρκινογενείς και ε, τις ε, ουσίες που προκαλούν αλλοιώσεις. Πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία αυτή επιγόντως. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα προκειμένου να προσαρμόσουμε καλύτερα τις συνθήκες εργασίας όσων πάσχουν από καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Θα ζητήσω επίσης από την Επιτροπή Μελέτη Αντικτύπου για τους ενδεχόμενου κινδύνους των ανατεχνολογιών στον τόπο εργασία συγκεκριμένα. Και τέλο. θα ήθελα μια σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κατάλογο των επαγγελματικών ιστανιών να την δούμε να μετατρέπεται πλέον σε οδηγία. Σήμερα χρειάζεται επικαιροποίηση του καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών που αυτή η σύσταση. Συνάδελφοι, η έκθεση αυτή θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο κάνοντας πολύ θόρυβο. Διότι θα πρέπει το ανθρώπινο όνειρο εργαζόμενοι να μπουν στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών εργασίας. Uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Ράπτη τώρα. Παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Εκ αρχής να ευχαριστήσω την κυρία Νταλίλη Κροσμπάχ και να την συγχαρώ για τους πολύ φιλοδοξούς στόχους που έχει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπερογνώμονες για τις πολλές πληροφορίες που μας έδωσαν με πολλά στοιχεία, στατιστικά στοιχεία, πολύ αξιόλογες συμβολές που θα εκμεταλλευτούμε γιατί χωρίς αυτά τα στατιστικά στοιχεία και τα εκδημητικά στοιχεία δεν μπορούμε να εκπονήσουμε μια πολιτική. Θα περισσώσει τρία σημεία καταρχήν. Αυτά τα, αυτές οι, οι συμβάσεις ε, αυτό αυξάνεται όσο πάει περισσότερο λόγω της κρίσης και βέβαια έτσι υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, που οδηγούν σε δυστυχήματα. Τα 168.000 θύματα ε, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό ο ρυθμός και θα πρέπει να έχουμε ένα όρμα μηδέν, όπως για, τις, για τους θανάτους στις οδικές μεταφορές και θα πρέπει να ελέγχεται πολύ περισσότερο η παράνομη εργασία, γιατί η παράνομη εργασία οδηγεί σε πίεση και η πίεση οδηγεί σε δυστυχήματα. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στις δημογραφικές αλλαγές. Δημογραφικές αλλαγές. Η... Το προσδόκιμο ζωής ε, του πληθυσμού αυξάνεται. Καλό είναι. Το χαιρετίζουμε γενικά. Αλλά λόγω της ε, πίεσης στα συστήματα στακτοδόσης είναι αναγκασμένος ο εργαζόμενος να παραμείνει περισσότερο στην εργασία του. Και αυτό δεν είναι πάλι εύκολο όταν περνάνε τα χρόνια και οδηγεί σε μια ανασφάλεια που οδηγεί πάλι σε ατυχήματα. Νομίζω η διαβίου μάθηση εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι όσο πάει και περισσότερο σημαντική στο μέλλον γιατί σε ορισμένες θέσεις απασχόλησης είναι αδύνατο να εργαστεί κανένας μετά τα 60 και θα πρέπει να μπορεί να έχει μια πιο ελαφρά εργασία και για να την πετύχει αυτή θα πρέπει να έχει μια νέα κατάρτιση. Τρίτον, θα ήθελα να αναφέρω αυτές τις νέες μορφές εργασίες, ιδίως στο τομέα της υγείας αυτό με όλα αυτέ τι χημικέ ουσίες, παραδείγματο χάρη στα καθαριστήρια ή και τις νέε τεχνολογίες και όλα αυτά που σχετίζονται με ακτινοβολίε και όσε αυτέ τι ψυχοσωματικές ε, ασθένειε που αυξάνονται και που θα πρέπει να βρούμε και για αυτές απαντήσεις. Ε, έχει προχωρήσει η ώρα και άλλοι θα θέλουν τον λόγο, γι' αυτό δεν θα αναπτύξω περισσότερο το θέμα μου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ράπτη και μετά ο κύριος Χέσου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι, είμαι εξαιρετικά ευτυχής που μπορώ να δηλώσω ότι βρίσκομαι στην ίδια κατεύθυνση με την εισηγήτρια. Ε, ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε το θέμα ε, με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι θα είναι πολύ λιγότερη η δική μου δουλειά. Ε, Ωστόσο, θέλω να τονίσω μερικά πράγματα. Θα ξεκινήσω από τον τομέα του στρες και του άγχους, που μας ανέπτυξε ιδιαίτερα ο τελευταίος ομιλητής. Συμφωνώ απολύτως και θα πω το εξής. 14 με 17 Ιουλίου πρόκειται να γίνει στην Ικαρία, ένα ελληνικό νησί, ένα συνέδριο. Το συνέδριο αυτό θα εξετάσει το γιατί ζουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες οι Ικαριώτες, οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Η απάντηση είναι ότι ζουν περισσότερο διότι αντιμετωπίζουν την εργασία τους και τον τρόπο ζωής τους με το λιγότερο δυνατό στρες. Επίσης, ένας δεύτερος λόγος είναι η διατροφή τους. Το αναφέρω αυτό γιατί θεωρώ ότι έχει άμεση σχέση με τον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας. Το στρες παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην Ευρώπη πάνω από 90 χρόνια ζει το 0,1% του πληθυσμού. Σε αυτό το μικρό ελληνικό νησί στην Ικαρία το ποσοστό αυτό είναι δεκαπλάσιο. Αυτό επιβεβαιώνει πλήρως τα όσα ακούστηκαν προηγουμένως σε σχέση με την επίπτωση του στρες, του άγχους στον τομέα της εργασίας. Είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ένα κομμάτι του στρες οφείλεται σε αυτό που υπόθηκε σε αυτή την αίθουσα, στο ότι στον ίδιο χώρο εργασίας μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους με δύο, τρεις ή τέσσερις διαφορετικές συμβάσεις. Ένας εργαζόμενος έχει σχέση αορίστου χρόνου. Άλλος εργαζόμενος έχει σχέση ορισμένου χρόνου, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Ένας τρίτος εργαζόμενος είναι μεταφερόμενος εργαζόμενος από άλλο κράτος. Έχει πρόβλημα με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, έχει πρόβλημα με τον τρόπο της ασφαλιστικής του κάλυψης. Άλλα ζητήματα. Ξεκινώ από την πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Η πρόληψη έχει να κάνει με την ενημέρωση και με διάφορους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως το διαδίκτυο. Η ενημέρωση πρέπει να αφορά κατά τη γνώμη μου και τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρομεσαίες, τους νέους και τους γυρεότερους. Τους νέους για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Πρώτον, διότι συνήθως οι νέοι απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και δεύτερον, γιατί οι νέοι υπερτιμούν τις δυνάμεις τους και υποτιμούν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Όσον αφορά την ενημέρωση των γυρεότερων, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την κατάρτιση που χρειάζονται, όπως είπε και ο συνάδελφος, αλλά και με το γεγονός ότι πρέπει να ενημερώνονται για τους νέους τύπους κινδύνων που φέρνει η εξέλιξη της τεχνολογίας σε κάθε εργασία. Η επανάληψη της κατάρτισης είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Και εδώ θεωρώ ε, πραγματικά αναγκαίο να πω ένα μικρό παράδειγμα από μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση που έχει ένα υποκατάστημα σε μία πόλη στο βορρά της Ελλάδας. Δεν θα αναφέρω το όνομα για να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση ή δυσφήμιση. Ε, η εταιρεία αυτή κατασκευάζει ρούχα. Στα ρούχα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο έλεγχος των χρωμάτων. Έτσι λοιπόν υπήρχε μία ομάδα γυναικών, 15 γυναίκες, οι οποίες είχαν δουλειά τους να ελέγχουν το χρώμα. Μετά από κάποια χρόνια άρχισαν να υπάρχουν παράπονα στην επιχείρηση ότι το χρώμα από το μανίκι της μπλούζας δεν τέριαζε με το χρώμα της κυρίως μπλούζας. Όμως ήταν οι ίδιες εργαζόμενες που με την ίδια επιμέλεια έκαναν τη δουλειά τους. Αναστατώθηκε ο χώρος εργασίας, έψαχναν να δουν τι γίνεται. Ήταν πάρα πολύ απλό. Οι γυναίκες αυτές όταν ξεκίνησαν να κάνουν τη δουλειά ήταν 25 χρονών. Όταν εκδηλώθηκαν τα παράπονα ήταν 40. Τα μάτια τους δεν είχαν πια την ίδια δύναμη. Εκεί λοιπόν καταλάβανε πόσο, πόση σημασία έχει η συνεχής ενημέρωση αλλά και η κατάρτιση του δυναμικού. Διότι αυτές οι γυναίκες έφυγαν από τη συγκεκριμένη δουλειά, έπρεπε να καταρτιστούν να πάνε σε μία άλλη και νέες εργαζόμενες μικρότερης ηλικίας με μεγαλύτερη δυνατότητα στην όραση να μπουν στο συγκεκριμένο πόστο. Νομίζω ότι έχει σημασία να βλέπουμε πραγματικά ε, και παραδείγματα από το χώρο εργασίας. Η, χρηματο... η κατάρτιση βέβαια χρειάζεται χρηματοδότηση. Και εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα κράτη-μέλη που πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα και μία ιδέα είναι ότι μπορούμε ε, να, να στηρίξουμε οικονομικά αυτή την προσπάθεια όχι μόνον μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά προτείνω και μέσα από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Γιατί μιλάμε για πρωτοποριακές έρευνες, για νέες πρακτικές και για καλύτερη εφαρμογή ε, κανόνων στην ασφάλεια της εργασίας όταν μπαίνει και η καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξέρω ο χρόνος κυρία Πρόεδρε, τελειώνω, ε, ε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξέρουμε όλοι ότι αντιμετωπίζουν ε, το ζήτημα της χρηματοδότησης και του κόστους. Άρα θα πρέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τις συνδράμουμε. Θεωρώ επίσης ότι σε αυτήν την στο αντικείμενο αυτής της έκθεσης που ε, ετοιμάζει η συνάδελφος ε, Νταλή έχει, να κάνει, έχει με πολύ μεγάλη σημασία η συνεργασία και ο συντονισμός όλων αυτών των, ε, πώς να το πω, των ευρωπαϊκών οργανισμών που εργάζονται για την ασφάλεια και την υγεία της εργασίας και που είχαμε την τιμή σήμερα να σας έχουμε εδώ να μας δώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Ο συντονισμός μεταξύ σας έχει τεράστια σημασία. Ε, νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε κανόνες, να έχουμε έλεγχο των κανόνων εάν εφαρμόζονται και αν δεν εφαρμόζονται να υπάρχει ε, ε, ε έρευνα γιατί δεν εφαρμόζονται. Πρέπει επίσης κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις που να τις κάνουν να θέλουν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια. Και από την άλλη μεριά να υπάρχουν ποινές αλλά και επιβράβευση των επιχειρήσεων. Αυτά είναι ε, συνολικά τα ζητήματα που εγώ ήθελα να θέσω στον χρόνο που έχουμε και ε, ένα τελευταίο σημείο είναι το εξή. Αισθάνομαι την ανάγκη να το υπογραμμίσω. Ε, το Eurofound, οι οργανισμοί από τους οποίους εκπροσωπείται και κάνουν εξαιρετική δουλειά κατά τη γνώμη μου, σήμερα σε αυτήν εδώ τη συζήτηση ε, έδωσαν, την ευκαιρία, έδωσαν την απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν το έργο τους και την αποτελεσματικότητά τους. Το λέω αυτό γιατί πριν δύο ή τρεις ολομέλειες στο Στρασβούργο ετέθη για μια ακόμη φορά το θέμα της χρηματοδότησης των οργανισμών αυτών και αν πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, να μην υπάρχουν ή να συγχωνευτούν. Ε, επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και τότε, θεωρώ ότι οι οργανισμοί αυτοί είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, μας βοηθούν να κάνουν τη δουλειά μας και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Uh, Mrs. Hirsch, followed by, uh, Κυρία Χίρς. Okay. Σας παρακαλώ στο δυνατόν πιο σύντομα, διότι πρέπει να μιλήσουν και οι εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα Έχω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις να κάνω για το θέμα, αλλά σήμερα εκπροσωπώ τον σκιώδη συγητή της ΑΝΤΕ, ε, τον κύριο Κρόιτσμαν, και θα περιοριστώ στα δικά του σχόλια. Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τους φιλελεύθερους και χαιρετίζουμε βέβαια γρητά το γεγονός ότι η Κομισιόν ε, έχει υποβάλει αυτή την ενδιάμεση μεθόδου Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία. Ο κ. Κρότ σημειώνει ότι έχουν γίνει πολλά ήδη και έχει έρθει για συνεργασία με την εισηγήτρια. Ε, βλέπουμε όμω επίση ξεκάθαρα ότι πολλά πρέπει να γίνουν σε αυτό το τομέα. Επίση, θα ήθελε ο κ. Κρότσμα να αναφέρει ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν εσωτερικές διατάξεις που ξεπερνάνε μάλιστα τις ε, κρατικές ε, διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων και δίνει το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου σήμερα ένα μεγάλο τμήμα των δυστυχημάτων ε, εξετάζονται από την κρατική από την κρατική οργάνωση ασφάλισης ατυχημάτων όσον αφορά τους τα ατυχήματα στο καθοδόν προς από την εργασία για τα οποία ο εργοδότης δεν έχει καμία επίδραση. Επίσης, ο κύριος Κρόσμαν ε, θεωρεί ότι δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικά πολλές διατάξεις για την προστασία της υγείας. Κάθε εργοδότης ξέρει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η υγεία των ε, συνεργατών του. Γιατί αν εργαζόμενος αρρωστήσει, ε, επιβαρύνεται η επιχείρηση. και γι' αυτό έχει ένα ίδιο συμφέρον, ιδίω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να εγγυάται ο εργοδότης μια υγιή θέση απασχόλησης. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΜΜΕ είναι εκείνες οι οποίες δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης και που επιβεβαιώνονται με τις περισσότερες διατάξεις. Ενώ μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν πιο εύκολα να πληρούν τις ε, νομοθετική αυτές διατάξεις. Γι' αυτό υποστηρίζει ο κ. Κρότσμαν την ιδέα τη ομάδα εργασία για την μείωση τη γραφειοκρατία που αναφέρεται στο έγγραφο εργασία και να εξαιρεθούν μικρέ εταιρείε σε τομεί που δεν φέρουν ιδιαίτερα ποσοστά κινδύνου. Και θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον την έκθεση της κυρίας Ντέλη και χαίρεται για μια καλή συνεργασία μαζί της. Ευχαριστώ κύριε Σπαρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές και προγράμματα από τις διάφορες υπηρεσίες για την ποιότητα των ε, ομιλιών τους και των σκέψεων που μας παρουσιάσαν. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι χάρηκα ακούγοντας αυτά που είχε να μας πει η συγγητριά μας η Καρή Μαντελή για τους προσανατολισμούς που θα δώσει στην έκθεσή της που από ό,τι μας είπε είναι πραγματικά αρκετά πλήρης και φιλόδοξη και θα μπορούμε έτσι να δούμε την κοινή μας θέση για να έχουμε κοινά σχέδια που θα στεφτούν από επιτυχία. Οπωσδήποτε ξέρουμε ότι το να ζει κανένας στις νήσους της Ελλάδας ε, εγγυάται μακροζωία. Απ' την άλλη μεριά βέβαια η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ε, περιγράφτηκαν όλες οι δυνατότητες ε, ασθενειών στον τόπο και προς το τέλος μάλιστα αναφέρθηκαν και τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν έξω από τα εργονομικά προβλήματα και προβλήματα εκθέσεως σε κάποιες ουσίες και η πρόληψη αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να γίνεται με διάφορες ε, παραμένες, δηλαδή υπάρχει ο εργοδότη που θα πρέπει να συμβάλλει τόσο ώστε να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στα μέσα που τους διαθέτει. Θα πρέπει επίσης να παρεμβαίνουν οι κοινωνικοί εταίροι, θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση πρώτη σημασία η ε, ιατρική εργασία και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, που δεν έχουν ποτέ πρόσβαση σε αυτή την ε, ιατρική. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί σε επιχειρήσεις των οποίων εργαζόμενων δεν έχουν πρόσβαση στου γιατρούς εργασία ούτε προληπτικά ούτε ε, κατόπιν κάποιων προβλημάτων. Υπάρχει επίση ένα άλλο σημαντικό σημείο η σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της, έργας, της ε, ιατρικής εργασίας και των ανθρωπίνων πόρων, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη του στρες, ε, του άγχους. Ε, επίσης, η επαγγελματική κατάρτιση ή επανακατάρτιση σε περίπτωση δυστυχήματος ή εξελιξη ανητικής του εργαζομένου όσον αφορά την αρρώστια του παραδείγματο κάνει δυστύχημα, ασθένεια ή ακόμα και εγκυμοσύνη για μια γυναίκα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα νέο προσανατολισμό, προσωρινό ή μόνιμο. Και αυτή η εταιρική σχέση θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ανθρωπίνων πόρων και τη ε, ιατρική εργασία. Θα ήθελα επίση να πω ότι πολλέ φορέ επιχειρήσει, σε ορισμένε χώρε τουλάχιστον, Υπάρχουν ορισμένε επιχειρήσει που έχουν υψηλά επίπεδα δυστυχημάτων και γι' αυτό υπόκεινται σε καιρό. Θα πρέπει λοιπόν να διδοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για να α, μειώσουν τα προβλήματα, τα δυστυχήματα αυτά, ίσως με κάποια οικονομικά κίνητρα. Ε, όλα αυτά νομίζω ότι είναι σύμφωνα με τις σκέψεις που κάναμε και πάνω σε άλλες εκθέσεις όπως η κινητικότητα των εργαζομένων και την αποσπασία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοική ισχύρενση, ε, άτομα με ειδικές ενάγκες στον τόπο εργασία. Και η τελευταία αναλύση είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε μεταξύ των κρατών μελών κάποια κατά κοινή νομοθεσία για την ε, σκοπιά αυτή της ε, πρόληψης των προβλημάτων τόπου εργασία είτε φυσικών είτε ε, ψυχολογικών. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία που πέρασαν στη διάρκεια των ετών εφαρμόζονται και μεταφέρονται σε κάθε κράτος μέλος. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιώδες για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, διότι αν δεν εφαρμόζονται ε, υπάρχουν προβλήματα και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει διαδικασίες επί παραβάση για τα κράτη-μέλη που δεν τα εφαρμόζουν και ως Επιτροπή πρέπει να ελέγχουμε. Να πω και κάτι για τους προσωρινά απασχολούμενους. Ε, συμφωνώ σε κάποιο βαθμό με αυτά που είπαμε ε, οι συνάδελφοι. Ε, εάν η προσωρινή εργασία ε, δεν είναι επιλογή κάποιου ανθρώπου. Κάποιοι όμως επιλέγουν να εργάζονται με προσωρινή απασχόληση. Αυτό δεν νομίζω ότι επιδεινώνει τα επίπεδα άγχους. Αν έχουν τη δυνατότητα επιλογής, για παράδειγμα. Αν κάποιος όμως αντί για πλήρη απασχόληση του δίνεται σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, τότε σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κάποιοι το επιλέγουν λόγω χρονικών περιορισμών, λόγω συγκεκριμένου τρόπου ζωής τους. Ε, όσον αφορά τώρα το άγχος, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ικαρία διότι νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας για να μειώσουμε τα επίπεδα του άγχους μας. Σημείωσα αυτά που ακούσαμε για το στρες, ε, δεν γίνεται αρκετή έρευνα για το άγχος και είναι πολύ δύσκολο να δούμε κατά πόσον ε, οφείλεται στο χώρο εργασίας, αν είναι απλώς συνσωρευμένο άγχος και πώς μπορούμε να κρίνουμε για ποια μορφή μιλάμε. Πώς μπορούμε ότι κάποιοι έχουν περισσότερη τάση να αγχώνονται και κάποιοι άλλοι όχι. Θα πρέπει να γίνει και περισσότερη δουλειά για τα επίπεδα άγχους στο χώρο της εργασίας και νομίζω ότι οι οργανισμοί ε, θα μπορούσαν να το εξετάσουν ε, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, ώστε να διαπιστώσουν πώς συνεισφέρει το άγχος ε, σε αρκετούς άλλους παράγοντες. Βεβαίως, πόρα απέχουμε ακόμα από αυτό και θα πρέπει να εξετάζουμε και το άγχος για τις διάφορες οδηγίες που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Εάν όμως κάνουμε αυτή την εξέταση χωρίς να έχουμε στοιχεία, δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Καλό θα ήταν να περιμένουμε να έχουμε κάποιες ενδείξεις και να δουλέψουμε λίγο πιο επισταμένα για να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα του άγχους με τη, σε σχέση με την εργασία. Όλοι θεωρούμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να γίνει με πιο διεξοδικό τρόπο, ε, να μην κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις και να μην αγχώσουμε ε, όλες τις οδηγίες συμπεριλαμβάνοντας και το άγχος εκεί χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τα στοιχεία που χρειάζονται. Κυρία Αντελή, δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα έχετε το χρόνο τώρα, αλλά σίγουρα θα λάβετε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που ακούσατε, ε, τα όσα είπαν τα υπόλοιπα μέλη και θα έχουμε άρθρονο χώρο στη διάθεσή μας να το συζητήσουμε. Να δώσουμε δύο λεπτά στον κάθε ένα από τους ε, ειδικού μας. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας, θα είμαι πολύ αυστηρή Καταρχάς να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καμαρότα. Έχετε το λόγο. Ε. Πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω όλους για τις χρήσιμες συμβολές τους στην όλη συζήτηση για την δημιουργία ενός νέου πολιτικού πλαισίου στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας και υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ ε, είναι εκείνη που πρωτοστατεί στις πρωτοβουλίες αυτές, προφανώς έχει να μας δώσει και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ, αλλά ενδιαφέρεται το ίδιο και να μας ακούσει. Και κυρία Ντελή, ελπίζουμε ότι και σε εσά θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το έργο σας, αλλά ακούμε και όσα λέτε. Είναι πολλές οι ελλείψεις, τα κενά που θα πρέπει να καλύψουμε και κατά τα άλλα να σας επισημάνω μια αρχή στην οποία παραμένει πιστή η Επιτροπή μας. Ο Επίτροπος παραμένει πιστός στην αρχή της επικουρικότητας με το άρθρο 150 της συνθήκης. Αυτό προβλέπει για την Επιτροπή τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια σειρά πρωτοβουλειών και να, φυσικά και νομοθετικών. Βεβαίως κάποια στοιχεία ε, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο Επίτροπος λοιπόν στο μέλλον θέλει να αναζητήσει τον καταλληλότερο τρόπο να συντονίσουμε τις πρωτοβουλίες, τις ευρωπαϊκές με τις εθνικές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Τάκαλα. Ε, σχόλια. Πρώτα απ' όλα για τους προσωρινούς εργαζόμενους. Δεν είναι όλοι αναγκαστικά ευάλωτοι. Και κάποιοι φοιτητέ λόγου χάρη είναι πιο ευάλωτοι όταν εργάζονται ως ασκούμενοι. Εγώ έχω υπήρξει, υπάρξει μετανάστης ως εργαζόμενος για πάνω από 30 χρόνια και έχω εργαστεί σε εξαιρετικές συνθήκες, ακόμα και σήμερα. Αυτό ισχύει. Τέλος πάντων, το άγχος είναι κάτι Αλλά δεν είναι κάτι που σκεφτήκαμε για να κουράσουμε τους εργοδότες και να τους αναγκάσουμε να ασχοληθούν με κάτι καινούριο. Όχι. Είναι ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Και δημιουργεί, έχει ακριβώς και σοβαρές επιπτώσεις. Είναι μείζονο σημασία για την εργασία. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια αποτελέσματα πρέπει κατά να δούμε τους παράγοντες που συντελούν πολλοί ε, συνδυάζονται. Το άγχος, ο φόρτος εργασίας, ε, οι ευθύνες και η ανάληψη αποφάσεων Αυτά όλα επιτείνουν το έγχος, λόγω να, το άγχος. Λόγω διαρθρώσουν επίσης κάποιοι φεύγουν από τις επιχειρήσεις και αυτοί που μένουν λαμβάνουν ακόμη περισσότερες ευθύνες. Αυξάνονται οι πιθανότητές τους για καρδιαγγειακές παθήσεις. Το άγχος τους, αλλά και αυτοί που μένοντας στη δουλειά όπως έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους καρδιαγγειακής θνησιμότητας. Κάτι άλλο που μας ε, ικανοποιεί Ιδιαίτερο είναι ότι νομίζω ότι με όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε συλλέξει και με το ενδιαφέρον που δείχνετε θα έχετε μια εξαιρετικά φιλόδοξη έκθεση. Ευχαριστούμε. Η συζήτηση ήταν συναρπαστική για κάποιον που ασχολείται με την έρευνα. Διότι ο ερευνητή γνωρίζει ότι η γενίκευση δεν είναι στοιχείο της έρευνας. Πρέπει κανείς να πηγαίνει στις λεπτομέρειες για να μπορεί να εξειδικεύει τη σκέψη του και του συλλογισμού του και τα συμπεράσματά του. Αυτή η συζήτηση λοιπόν για μένα ήταν συνεργαστική. Μερικές σκέψεις για το άγχος. Στα γαλλικά προφανώς διότι ο τελευταίος ομιλητής υπό τη μακροζωία Μίλησε για τη μακροζωία λοιπόν στην Κρήτη. Η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Με πολλές λεπτομέρειες εξίσου περίπλοκες. Και προβάλλονται επιχειρήματα, πληθώρα επιχειρημάτων, εκτός επιχειρήσεων και εντός επιχειρήσεων. Όμως η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να μας κάνει να παραγνωρίσουμε τη σημασία του χώρου εργασίας. Είναι πολλές, ε, ο χώρος εργασίας μάλλον έχει τόσες πολλές προεκτάσεις και τόσους παράγοντες που αλληλεπιδρούν που δεν μπορούμε παρά να αναλάβουμε δράση. Υπάρχει μάλιστα μια νέα γενιά ερευνητών που λένε ότι την παρακολούθηση των προσπαθειών και την αποτίμησή του πρέπει να την αναλαμβάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι πώς, ε, πώς προχώρησαν τα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο, τι δείκτες χρησιμοποιήθηκαν ώστε να εκτιμηθεί πρόοδος σε εθνικό επίπεδο. Παρακαλούμε μπορείτε να κλείνετε. Ε, ναι. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπάρχει και το στοιχείο της επικουρικότητας εδώ. Και οπωσδήποτε ο χώρος εργασίας ε, πρέπει να διέπεται και από αυτήν την αρχή. Ευχαριστώ, αλλά αν ξεπεράσουμε το χρόνο μας και εγώ θα ξεπεράσω τα επίπεδα κοπόσεώς μου και άγχος μου. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες, όλους όσους συνεισέφεραν στην κουβέντα. Να πω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 16 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, συζήτηση για τις τροπολογίες 26 ε, Οκτωβρίου, 7 Νοεμβρίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή, και στην δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου η ολομέλεια θα εξετάσει το θέμα αυτό. Θα μπορέσουμε λοιπόν να το ξαναδούμε στην Επιτροπή μας και να το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερως. Επόμενη συνεδρίαση, στην επόμενη μάλλον... Η επόμενη συνεδρίαση μας προβλέπεται στις 8 Σεπτεμβρίου μόλις, θα χαρείτε όλοι ιδιαίτερως φαντάζομαι, στις 9 το πρωί. Καλές σας διακοπές λοιπόν, αν φέγετε για διακοπές, εάν μένετε στις εκλογικές σας περιφέρειες επίσης και δουλεύετε, μην αγχωθείτε. Σας ευχαριστούμε.